Bonjour, bonjour, monsieur, Nous Sont pas très nombreux, mais... Καλημέρα σα, κυρίε και κύριοι. Δεν είμαστε και πολύ με στην αίθουσα. Τραβάει. Θα αργήσουμε. Θα αρχίσουμε. Alors, oui, tout de suite, madame. D'abord, vous annoncez l'ordre du jour. Oui. 6 5. Porządek dzienny dzisiaj będzie nieco zmieniony, tak jak ustalaliśmy wczoraj, jako punkt pierwszy będzie punkt... Έχει τροποποιηθεί κατά τη ημερήσια διάταξη. Θα ασχοληθούμε πρώτα απ' όλα με το σημείο 26 για τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Μετά το 25, δηλαδή ΑΕΠ και πέρα από αυτό η μέτρηση πρόοδου σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο και μετά θα συνεχίσουμε κανονικά όπως προβλέπεται στην ημερήσια διάταξη. Παρουσία δηλαδή χαμηλών ποσοτήτων γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών στα τρόφιμα και κοινή γεωργική πολιτική. Πριν να αρχίσω, λέει ο πρόεδρο, θα ακούσουμε την κυρία Χάμς. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά που μας είπε ο Επίτροπος Oettinger χθες στην Επιτροπή μας και θα ήθελα να θέσω το ερώτημα και πάλι στους εκπροσώπους της Κομισιόν, ελπίζω ότι είναι εδώ παρόντες σήμερα, αλλά θα ήθελα να κάνω και μια αίτηση προς το Προεδρείο της Επιτροπής μας. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των γερμανικό τύπο, ιδίως στο περιοδικό Der Spiegel, μετά από την παρουσίαση του κυρίου ο δείκτης χρηματιστηρίου DAX έπεσε σημαντικά και σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης μια εκπρόσωπος του κυρίου Έτιγκερ μιλώντας προς τα μέσα ενημέρωσης είπε ότι οι αξιολογήσεις που ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης για τον κύριο Έτιγκερ είναι απλώς η εντυπώσεις που σχημάτισαν τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό με ενοχλεί. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο ο κύριος Σέτιγκερ είναι σε επαφή με την Ευρατόμ, με τον Φορέα Διεθνούς Ατομικής Ενέργειας και με τις ε, Εθνικές Υπηρεσίες Ατομικής Ενέργειας που όλες παρακολουθούν από πολύ κοντά και αξιολογούν τα γεγονότα στην Ιαπωνία. Θα ήθελα λοιπόν να έχω και μία θέση σε σχέση με αυτά που είπε η εκπρόσωπος του κυρίου Έτιγκερ, γιατί αυτό δεν νομίζω ότι είναι μία κατάσταση η οποία μπορεί να ευνοήσει την εμπιστοσύνη στον πληθυσμό. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Προεδρεύων. Προτού τώρα δώσω το λόγο σε άλλους συναδέλφους, θα ήθελα να σας πω ότι προχθές Ήμουν σε μια άλλη συνάντηση με τον Επίτροπο Έτιγκερ, όπου είπα ακριβώς τα ίδια πράγματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Με ταυτόσιμες ε, λέξεις. Τώρα δεν κατάλαβα γιατί τα μέσα ενημέρωση δεν αντέδρασαν τότε, ο κύριος Ζέμπερ. Σας ευχαριστώ. Έρχομαι και πάλι στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε πολλά σημεία στην ημερήσια διάταξη. Εγώ δεν βρήκα, βρήκα στην ημερήσια διάταξη το σημείο αυτό που ανέφερε η κυρία Χάμς επειδή έχουμε πολλά σημαντικά σημεία να εξετάσουμε σήμερα, θα ήθελα να ζητήσω από τον Πρόεδρο να παραμείνει στην ημερήσια διάταξη. Έχει νόημα το ερώτημα της κυρίας Χάρμς, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε εδώ τους εκπροσώπους της Κομισιόν, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για να κάνουμε μια συζήτηση για τα θέματα αυτά των δηλώσεων του κύριου Έτιγκερ και δεύτερον η ημερήσια διάταξη για την Επιτροπή μας έχει κανονιστεί εδώ και πολύ καιρό. Θα ήθελα λοιπόν να προχωρήσουμε γιατί δεν βλέπω να έχει γίνει κάποια αίτηση αλλαγή τη ημερησία διάταξη. Σα ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο. Ο κύριο Πρόντι, αν θέλει το λόγο. Αργότερα, αργότερα, ήταν για αργότερα η παρέμβαση που ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ. No tak, tylko że Ο συνάδελφος Πρόντι δεν θέλει να μιλήσει, αλλά άλλοι ζητούν το λόγο. Εγώ δεν θέλω να γίνει συζήτηση. Η κυρία Χάρμζα έκανε μια δήλωση, αλλά δεν είναι αυτή η υπόθεση. Ε, μιλάμε για τα καύσιμα και το ραδιο, ραδιενεργά απόβλητα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Λέω κύριε Το ραδιενεργό, το νομικό πλαίσιο για τα ραδιενεργά απόβλητα ε, μας απασχολεί εδώ πρόκειται για μια αναθεώρηση της ε, σχετικής οδηγίας του 2003. Επίσης ε, είναι η οδηγία 71-2009 που προστίθεται εδώ και ασχολείται με τη διαχείριση των πυρηνικών καυσίμων στους χώρους παραγωγής τους. Όποιο και αν είναι το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας, ε, θα πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα αυτό, γιατί προς το συμφέρον ε, της ασφάλειας, ε, τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια. Δεδομένων των χαρακτηριστικών αυτού του τύπου των αποβλήτων, πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η βασική αρχή Τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων είναι η αποθήκευσή τους και η απομάκρυνσή τους από τους ανθρώπους από τη στιγμή που είναι, ε, για όσο μάλλον χρόνο, είναι ραδιενεργά. Ωστόσο, σε περίπτωση αποβλήτων υψηλού επίπεδου ραδιενέργειας υπάρχει η επιστημονική βεβαιότητα πως η ταφή τους σε μέγα βάθος είναι η μόνη ασφαλής λύση. Όμως, στα κράτη-μέλη δεν υπάρχουν αρκετοί τέτοιου τύπου αποθηκευτικοί χώροι για υψηλού επίπεδου ραδιενεργά απόβλητα. Η πυρηνική ενέργεια χρησιμοποιείται εδώ και 50 χρόνια, όμως δεν υπάρχει κάποιος ε, τελικός ε, προορισμός ταφής η ευθύνη για τα απόβλητα και τα ραδιενεργά απόβλητα είναι βαραίνει τα κράτη-μέλη. Και εμείς θα πρέπει να αποφύγουμε να επιβάλλουμε τέτοιο ανεπιθύμητο φορτίο στις μελλοντικέ γενναίες. Η ευθύνη λοιπόν βαραίνει τις σημερινές γενναίες που έχουν ωφεληθεί από την πυρηνική ενέργεια και από την παραγωγή ηλεκτρισμού ε, και θα πρέπει εμείς να διαχειριστούμε τα πυρηνικά απόβλητα. Παρόλα αυτά, ε, ε, θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις σε σχέση με τη διαχείριση και την ε, ταφή αυτών των αποβλήτων. Γενικό στόχος της οδηγίας είναι να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων και των ραδιενεργών αποβλήτων προς το συμφέρον των μελλοντικών γενεών και έτσι ώστε να συνεχιστεί η χρήση αυτής της πυρηνικής τεχνολογίας για την ιατρική, την έρευνα και τη γεωργία καλούνται όλα τα κρατημέλη να αναλάβουν τις ε, κατάλληλες αποφάσεις ώστε να ε, εισάγουν τα κατάλληλα προγράμματα διαχείρισης ε, των αποβλήτων αυτών για τα αναλωμένα καύσιμα. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην συμμόρφωση προς την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ισχύουσα και μάλλον οι χρησιμοποιούμενες πρακτικές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της εξέτασης αυτής της οδηγίας. Θα πρέπει να γίνεται βιώσιμη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και είτε μας αρέσει είτε όχι. Η πυρηνική ενέργεια αυτή τη στιγμή παράγει το 30% της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ορισμένα κράτη φτάνει και στο 80% δεν θα πρέπει να γίνει καμιά ανακατάταξη των ε, χρησιμοποιούμενων αυτών αποβλήτων όπως τα ραδιοενεργά απόβλητα γιατί υπάρχει γενικά συνένεση μεταξύ των εμπειρογνωμόνων ότι η, ταφή των αποβλήτων αυτών είναι η καταλότερη μέθοδος για τα τα πιο επικίνδυνα στερεοποιημένα τέτοιου είδους καύσιμα. Χρειάζονται βεβαίως έρευνες. Η έρευνα και οι τεχνολογικές εξελίξεις θα πρέπει να στηριχθούν ε, οικονομικά και οι συμφωνίες για τις εξαγωγές τέτοιων αποβλήτων με διάφορες χώρες θα πρέπει να εξεταστούν ανά περίπτωση. Υπάρχουν ορισμένε ειδικέ ε, περιπτώσεις όπου τα κράτη-μέλη έχουν στην αναλώσιμα καύσιμα για επανεπεξεργασία σε μη κοινοτικέ χώρε και ορισμένα από τα απόβλητα αυτής της κατεργασία παραμένουν στη χώρα υποδοχή. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούν να στέλνονται τέτοια απόβλητα πίσω στις χώρες όπου αρχικά ε, δημιουργήθηκαν αυτά τα απόβλητα. Ορισμένε τώρα περιπτώσεις, ε, ε, μάλλον οι περιπτώσει ασφάλεια δεν πρέπει να αναφέρονται αυτή την οδηγία. Είμαι πεπισμένο ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πολιτική στα κράτη-μέλη, η διαχείριση των ε, ραδιενεργών αποβλήτων είναι ένα επίκαιρο θέμα που πρέπει να λυθεί. Εδώ βέβαια μιλάμε για τεχνικά θέματα, θα πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την οδηγία σε ένα πολιτικό πεδίο μάχης για το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος, κύριε Πότς. Ποιος θα θέλει να λάβει το λόγο. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Κύριε Σπατολότσι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορεί κανείς να μην αναφερθεί και στη σημερινή σοβαρή διεθνή κατάσταση όταν μιλά για τέτοια θέματα που μας επιβάλλει να εξετάσουμε αυτό το τόσο λεπτό και σημαντικό ζήτημα με μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης. Χωρίς ωστόσο να αφήσουμε να παρασυρθούμε από δημαγωγικές, δημαγωγικά επιχειρήματα. Θα πρέπει συγκεκριμένα να προσεγγίσουμε το θέμα. Σε αυτή τη γραμμή εντάσσεται θετικά ο στόχος που βρίσκεται στη βάση αυτής της πρότασης οδηγίας που είναι να ορίσει έναν αρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για το, σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα. Η οδηγία εντάσσεται στο σύνολο των διεθνών ε, κανόνων και των κοινοτικών κανόνων για το θέμα αυτό. Η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι αρμόδια για το θέμα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τη συνθήκη Ευρατόμ. Μια κατάλληλη κοινοτική πολιτική, λοιπόν, θα έπρεπε να εγγυάται την απόλυτη προτεραιότητα της ασφάλειας των πολιτών και του σεβασμού του περιβάλλοντος. Με αυτούς ε, τους στόχους, μια ξεκάθαρη ευρωπαϊκή οδηγία που να είναι σωστά ε, διαρθρωμένη, διαφανής ε, και δεσμευτική και που θα ορίζει όλες τις βάσεις διαχείρισης από την αποθήκευση στην επεξεργασία μέχρι και την ταφή θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και ακριβώς απαιτείται ένα τέτοιο είδος ρυθμιστικού πλαισίου κυρίως όσον αφορά την ε, ταφή γιατί πολλές χώρες έχουν υπογράψει την κοινή σύμβαση της Διεθνούς Υπηρεσίας για την Ατομική Ενέργεια, αλλά δεν υπάρχει στην ουσία ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική μια τέτοια προσέγγιση, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν εθνικά προγράμματα για τη διαχείριση των ε, αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, με βάση την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που θα αφήνει χώρο και σε μορφές περιφερειακής κοινοτική συνεργασίας αλλά και εξωκοινοτικής συνεργασίας. Όλα με διαφάνεια όμως και ασφάλεια. Θα πρέπει επίσης να εγγυηθούμε υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας που θα συμμορφώνονται με τα όσα περιλαμβάνονται στις προηγούμενες οδηγίες της Ευρατόμου. E Ευχαριστούμε τον κύριο Μπερτολότσι. Η Άννα Ρόσπαχ τώρα για τη συντηρητική ομάδα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω τα εξαιρετικά σχόλια του κύριου Πότς και των λοιπόν συναδέλφων. Θα ήθελα μόνο να πω ότι πριν από ένα μήνα περίπου ήμουν ε, στη Φινλανδία και επισκέφτηκα ένα πυρηνικό εργοστάσιο και άρχισα να προβληματίζομαι για αυτό το θέμα. Γιατί θέλουμε να αποθηκεύουμε υπογείως τα απόβλητα αυτά, δεδομένου του ότι τα υλικά αυτά έχουν την μισή περίπου ε, από την αρχική τους ενέργεια. Πρώτα πρέπει να αποθηκευτούν σε υδάτινο περιβάλλον για 30 χρόνια πριν μπορέσουν να ε, αποθηκευθούν ε, υπογείως. Πρέπει να απελευθερωθεί δηλαδή μεγάλο κομμάτι από την αρχική τους ενέργεια προτού καν αρχίσουμε να συζητούμε την τελική διάθεση των αποβλήτων. Βέβαια ξέρετε πόσο σχολαστική είναι οι Φινλανδοί, τα κάνουν τα πράγματα όπως πρέπει και είδα ότι κάνανε γεωτρήσεις ε, και ρίχνανε κάψουλες ε, με τσιμέντο, ε, κάψουλες που περιείχαν τα απόβλητα αυτά. Η ενέργεια είναι τόσο μεγάλη που αν αποθηκευτεί ουσιαστικά δεν χρησιμοποιείται ενώ θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε στον τομέα της ιατρικής ή σε κάποιον άλλο τομέα. Ε, αποθηκεύονται αυτά τα απόβλητα σε κάποιες μεγάλες, πώς να τις πω, σουπιέρες ε, μέσα σε νερό για 30 χρόνια. Γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το υλικό εφόσον ακόμη περιέχει ενέργεια. Ευχαριστούμε κυρία Ροσμπα Ρεμπέκα Χάρμς. <clears throat> Ähm, ναι, και πάλι παίρνω το λόγο τώρα θα ήθελα να σταθώ στο θέμα που μας απασχολεί στην Επιτροπή μας. Στην Επιτροπή Βιομηχανίας ξεκινήσαμε την εξέταση της ε, πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το πρώτο το οποίο θα θέλω να πω ότι μου δημιουργήσε εντύπωση είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά με την, ε, μεταξύ της τρέχουσας επεξεργασίας και της επεξεργασίας της προηγούμενης οδηγίας. Αυτό ήταν μια πρόταση της Λοϊόλα για την τελική εναπόθεση των πυρηνικών αποβλήτων στην Ευρώπη. Τότε ο στόχος της οδηγίας αυτής ήταν να καταλήξουμε και σε μια σαφέστερη αντιμετώπιση για το πώς θα λάβουμε όχι μονάχα λύσεις για την εναπόθεση των αποβλήτων, αλλά να σκεφτούμε και τι θα κάνουμε με τα περαιτέρω πυρηνικά εργοστάσια που εσμένες στοχεύουν να δημιουργήσουν. Επομένως, όχι μονάχα να παραμείνουμε στα, στην απόθεση των ε, αποβλήτων, αλλά να είναι προϋπόθεση η τελική αναπόθεση των αποβλήτων προτού ξεκινήσουμε να έχουμε νέα πυρηνικά εργοστάσια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μου πολιτική ομάδα και επομένως η Επιτροπή Βιομηχανίας ε, θα πρέπει να γνωρίζει τις δυσκολίες οι οποίες παρουσιάστηκαν στην ε, Σουηδία για τους σταθμούς εναπόθεσης. Επίσης τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν σε ένα σταθμό εναπόθεσης ε, αναλωμένων ραδιενεργών υλικών στην Γερμανία. Εγώ έχω πει στην Επιτροπή μας ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να πάτε στην ε, Γερμανία και να, βρείτε, δείτε αυτό τον σταθμό πυρηνικών αποβλήτων όπου θα μπορέσετε πραγματικά να διαπιστώσετε και με τα ίδια σας τα μάτια τις δυσκολίες οι οποίες προκύπτουν όταν υπάρξει ένα πρόβλημα σε κάποιο σταθμό εναπόθεσης αποβλήτων. Παρ' όλα αυτά κανένας εισηγητής δεν αποφάσισε να πάει στη Χάσα, στη Γερμανία, να τα δει όλα αυτά. Τώρα για την πρόταση ε, οδηγίας θα ήθελα καταρχήν να παρατηρήσω ότι ο ορισμός των πυρηνικών αποβλήτων κατά τη δική μας άποψη δεν είναι ο σωστός ορισμός. Κάθε κράτος μέλος έχει την ελευθερία να αποφασίσει τι ακριβώς <clears throat> αποτελεί ε, ραδιενεργό απόβλητο. Ένα κράτος μέλος μπορεί παραδείγματος να χρησιμοποιήσει τα αναλωμένα καύσιμα ως νέα πρώτη ύλη για επανεπεξεργασία ή αλλιώς ως απόβλητα. Αυτό είναι κάτι το πολύ επικίνδυνο. Γίνεται δυνατό λοιπόν να προωθηθεί και η εξαγωγή των προϊόντων αυτών, των αναλωμένων καυσίμων σε τρίτες χώρες, γιατί αν δεν καθοριστούν, αν δεν θεωρηθούν ότι είναι απόβλητα, υπάρχει δυνατότητα ως προϊόντα επεξεργασίας να αποσταλούν σε άλλες χώρες και μιλάμε για προϊόντα τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα, όχι μόνο στη Ρωσία αποστέλλονται, αλλά και σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εξαχθούν. Επομένως, η πιο σημαντική διεκδίκηση της ομάδας μου για την περαιτέρω <clears throat> διαβούλευση που αφορά αυτή την οδηγία είναι η εξή. Αυτό το οποίο εμεί θέλουμε είναι η οδηγία αυτή να χαρακτηρίζει όλα τα ραδιοναργά απόβλητα ως απόβλητα, να τα καλύπτει όλα και όχι ένα μικρό τμήμα της μονάχα. Θέλουμε ότι αυτά τα οποία ε, είναι απόβλητα από την ανάκτηση ουρανίου να θεωρούνται πράγματι ότι είναι απόβλητα και επίσης τα απόβλητα τα οποία χρησιμοποιούνται τα οποία προέκυψαν μάλλον σε προηγούμενες χώρες από στρατιωτικές διαδικασίες, να θεωρηθούν επίσης απόβλητα. Όλα τα αναλωμένα καύσιμα θα πρέπει να θεωρούνται απόβλητα λοιπόν και επίσης οι εκπομπές ραδιενέργειας οι οποίες εκλείονται στο περιβάλλον, παραδείγματος χάρη στην ε, Λαχάγκ, στο σταθμό επανεπεξεργασίας αναλωμένων καυσίμων στην ε, Γαλλία, να θεωρηθούν ως ε, αντιμετώπιση αποβλήτων, γιατί δεν μπορεί κανείς να ελέγξει την ε, ραδιενέργεια η οποία εκπέμπεται από αυτούς τους σταθμούς. Και χωρίς την παρουσία τέτοιων μονάδων επανεπεξεργασίας δεν θα μπορούσαν οι βιομηχανίες ελαφρά την καρδία να δίνουν κάπου αλλού τα αποβλητά τους. Πρέπει λοιπόν να έχουμε επίσης τη δυνατότητα να έχουμε και μια <clears throat> καλύτερη και επακριβή μέτρηση Τη ακτινοβολία που εκλείεται από σταθμού, οι οποίοι είναι εκτός λειτουργίας. Αυτό είναι πράγματι σε μια πρακτική πολλών χωρών οι οποίες ε, παίρνουν πράγματι χαμηλής ραδιενέργειας υλικά και τα ενσωματώνουν παραδείγματος χάρη στην άσφαλτο των ε, αυτοκινητοδρόμων. Αυτό είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μου επέχει κινδύνους. Εμείς θέλουμε να αντιμετωπιστούν τα ιστορικά απόβλητα πρώτα απ' όλα με επαρκή τρόπο και η οδηγία αυτή, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει και μεγάλη επικαιρότητα, να την αντιμετωπίσουμε με ένα νέο πνεύμα και να λάβουμε υπόψη σοβαρά όλα τα προβλήματα τα οποία τίθενται από πιθανούς σεισμούς, όχι μονάχα για ατομικούς σταθμούς, αλλά και για σταθμούς εναπόθεσης αναλωμένων καυσίμων στην Ιαπωνία μετά από τον σεισμό υπήρξαν τεράστια προβλήματα ε, σε σταθμούς εναπόθεσης, προσωρινής εναπόθεσης ε, καυσίμων, ακόμα και σε σταθμό τελικής εναπόθεσης υπήρξαν προβλήματα λόγω του σεισμού, επομένως όλα αυτά πρέπει να, να επανεξεταστούν στο φως των εμπειριών που έχουμε τώρα συλλέξει. Επομένως, σε σχέση με την οδηγία, θα πρέπει να υπάρξει και μεγαλύτερη σαφήνεια για το ποιος είναι υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων και ποια θα πρέπει να είναι και η έκταση των διαβουλεύσεων με τους εμπειρογνώμονες σε σχέση με τη λήψη απόφασης. Δεν θεωρούμε ότι είναι σωστό να μείνουν αυτά τα θέματα απόλυτα ανοιχτά. Επίσης δεν μας φαίνεται ορθό να μείνει ασαφής η έννοια ότι τελικά ο παραγωγός είναι αυτός ο οποίος έχει την τελική ευθύνη για την τελική εναπόθεση και θέση σε ασφάλεια των ραδιενεργών υλικών. Δηλαδή η πραγματοποίηση και η υλοποίηση της αρχής ορυπαίνων ε, πληρώνει. Θεωρούμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μία αδυναμία της ε, τρέχουσας οδηγίας. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, χρηματοδοτικά μέσα για την τελική εναπόθεση μετά από 50 χρόνια δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη από τις εταιρείες οι οποίες λειτουργούν τους πυρηνικού σταθμούς. Για μας αυτό είναι επίσης ένα κομβικό σημείο το οποίο τονίσαμε και στην Επιτροπή Βιομηχανίας και εξέφρασα εκεί τη λύπη μου για το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια πραγματική ανταλλαγή απόψεων που να έχει λάβει χώρα μεταξύ των εισηγητών της, των σχεδόν εισηγητών της ε, Επιτροπής μας. Ο εισηγητή μας δεν έχει βρει αρκετό χρόνο για τα θέματα αυτά. Θα ήταν χρήσιμο όμως να έχουμε επαφέ για να μπορέσει να γίνει σαφής η θέση όλων των μελών της Επιτροπής μας. E, σας ευχαριστούμε κυρία Χάρμς. Ήταν πληρέστατη η τοποθέτησή σας. Ο Chris Davis τώρα από τους φιλελεύθερους, ο Βιτόριο Πρόντι, η Ροβάνα Πλάμπ και μετά ο κύριος Πότς. Κρίς, ευχαριστώ πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον, ε, την Αντώνιο Παϊβανόβα Εύκολα μπορεί κάποιος να έχει συγκαταβατική στάση για τέτοια ζητήματα, στο μέτρο που δεν υπάρχουν προβλήματα, αγνοεί κάποιος το ενδεχόμενο να προκύψουν προβλήματα. Όταν βλέπουμε την κατάσταση στην Ιαπωνία και κάποιες από τις αποκαλύψεις σχετικά με τη διαχείριση των πυρηνικών εργοστασίων, επιβεβαιώνουν την ανησυχία μας πάνω από 50 χρόνια ε, λειτουργούν αυτές οι μονάδες χωρίς ε, να ανησυχεί κανείς και βλέπετε πόσο τρομακτικά αποδεικνύονται όλα αυτά τώρα. Ε, βλέπουμε τα κάψιμα που βρίσκονται στις δεξαμενές ε, και ε, διευρύνονται οι δεξαμενές ε, ούτως ώστε να μπαίνουν περισσότερες ε, ράβδοι από τον αρχικό σχεδιασμό και αυτές οι δεξαμενές οδήγησαν στις διαρροές και στο πρόβλημα. Τέλος πάντων, στην πυρηνική βιομηχανία χρειάζεται διαφάνεια, χρειάζεται αμερόληπτος ανεξάρτητος έλεγχος ε, και κάποιοι προτάσουν ε, το θέμα της επιχειρηματικής εμπιστευτικότητας, αλλά με αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Ιαπωνία και ενδέχεται να επιδεινωθεί η κατάσταση τις επόμενες ημέρες. Ε, αυτά υπονομεύουν την εμπιστοσύνη που υπάρχει για την πυρηνική βιομηχανία μέρα με τη μέρα. Χρειάζεται απόλυτη διαφάνεια, είτε μιλάμε ε, για την ε, λειτουργία των εργοστασίων, είτε για την αποθήκευση των αποβλήτων. Θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα της μεταφοράς τους τώρα. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπω και τη χώρα μου η μεταφορά των αποβλήτων ανάμεσα σε πυρηνικές μονάδες δεν νομίζω ε, εδώ και 50 χρόνια να έχει δημιουργήσει κάποιο ναι. πρόβλημα. Ε, ποια είναι η ιδέα, τα καύσιμα, τις δεράδους ε, των καυσίμων να τις απομακρύνουμε από την Ιαπωνία και να επανεπεξεργαστούν ε, κάποιοι όπως το Ηνωμένο Βασίλειο αυτά τα απόβλητα. Ε, βέβαια σε σεισμογενείς ε, περιοχές ε, γίνονται επικίνδυνα τα πράγματα και άλλο είναι να στέλνετε τα απόβλητα σε μια τέτοια χώρα άλλο να τα στέλνετε μέσω θαλασσίων οδών. Μην ξεχνάτε ότι τα σκάφη βουλιάζουν, συμβαίνουν ατυχήματα. Τώρα, η μακροχρόνια αποθήκευση των αποβλήτων, άλλο ένα δύσκολο θέμα. Θα θέλαμε να ε, χρησιμοποιούνται βαθιά γεωλογικά στρώματα για την ταφή τους, αλλά ας μην ε, ε, ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα απόβλητα τόσο βαθιά μέσα στο έδαφος, κυρίως όταν είναι σεισμογενείς περιοχές. Πρέπει να υπάρχει μια διάταξη, μια πρόβλεψη, ώστε να μπορούμε να ανακτούμε αυτά τα απόβλητα οι επιστήμονες τελικά μάλλον θα βρουν ε, ε, τη λύση που μας υπόσχονται ε, εδώ και χρόνια ούτω ώστε με ασφάλεια να αποθηκεύουμε τα απόβλητα. Ας μην τα αφήσουμε σε, στην, σε υπόγειους χώρους ταφής, ας αφήσουμε τη δυνατότητα ανάκτησής τους από τις μελλοντικέ γενιές και ας μην τα θάβουμε και τα ξεχνάμε τα απόβλητα. Τώρα κάτι άλλο. Υπάρχουν συμβάσει ανάμεσα σε κυβερνήσει και πυρηνικά εργοστάσια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Ρωσία. Υπάρχει μια σύμβαση ανάμεσα στη Ρωσία και στη Βουλγαρία. Αν τώρα ε, νομοθετήσουμε και πάλι θα αναθεωρηθούν αυτές οι συμβάσεις ή λέμε απλώς ότι οι διατάξεις προβλέπουμε εμείς στην νομική πράξη καλύπτουν μόνο την επικράτεια της Ένωσης. Θα καλύπτουν και τα ραδιενεργά απόβλητα που έχουν παραχθεί, δημιουργηθεί μέσα στην Ένωση και έχουν εξαχθεί για επανεπεξεργασία. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντέιβις. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Εγώ πιστεύω πως θα έπρεπε αυτή να είναι μια ευκαιρία για μια ευρύτερη συζήτηση. Η Ευρωτόμα έκανε ωραία πράγματα όσον αφορά την ε, διοργάνωση της προστασίας από την αδενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά στην πράξη όλο αυτό το τμήμα, το πιο βιομηχανικό, στην ουσία καθορίζεται από το γεγονός ότι υπάρχουν δύο χώρες που έχουν πυρηνικούς εξοπλισμούς. Αυτό εμπόδισε να μπορέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναλάβουμε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την πυρηνική ενέργεια. Καλός ή κακός, αυτή είναι η υποθήκη που έχουν κληροδοτήσει η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρατόμ. Εμείς τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αν το πρόβλημα των αποβλήτων που υπάρχει θα πρέπει ε, να αντιμετωπιστεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συντονισμένη πρωτοβουλία ε, που δεν θα την αφήσουμε μόνο στα κράτη-μέλη γιατί πολύ συχνά δεν μπορούν μόνο τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Νομίζω πως είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή για να αποφασίσουμε τι είναι η Ευρατόμ, τι θέλουμε να κάνουμε με την Ευρατόμ, να κάνουμε πράγματα που πραγματικά να μετράνε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόντι, η κυρία Ροβάνα Πλάμπ και μετά ο κύριος Ζίμπερ που θα είναι και ο τελευταίος ομιλητής. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομο. Γιατί πολλά ε, Ήδη αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους. Καταρχήν υποστηρίζω τον κύριο Πότς. Αυτό που έχουμε όμως είναι μια πρόταση, πρόταση οδηγίας και εξάλλου είναι ένα πρόβλημα το οποίο βρίσκεται στην καυτή επικαιρότητα. Όχι μόνο τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην ε, Ιαπωνία, αλλά και μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ενδιαφέρει το θέμα των ενεργειακών υποδομών πριν και μετά από το 2020. Εξάλλου, σε σχέση με τη διαχείριση της οδηγίας αυτής και το σχέδιο έκθεσή μας, εγώ θέλω να αναφερθώ στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να τονίσω ότι εδώ δεν πρόκειται μονάχα για την διαχείριση σε ό,τι αφορά την προεπεξεργασία, επεξεργασία και την προετοιμασία για ενδιάμεση εναπόθεση. Δεν πρόκειται για αυτά. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια πλήρη παρακολούθηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων και να έχουμε και μια συντήρηση των χώρων όπου λαμβάνει η χώρα η προσωρινή αναπόθεση ή η οριστική αναπόθεση των πυρηνικών αποβλήτων. Εγώ συμφωνώ ότι εδώ η ευθύνη θα πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών, αλλά συγχρόνω μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί να υπάρχει και μια συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο και να υπάρξει και ένα συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι πολλέ φορέ τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο. Ο Ρίχα Τσέμπερ. Σα ευχαριστώ, πρόεδρε. Εμείς κατανοούμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να ασχοληθούν με τα θέματα της, ε, των ενεργειακών φορέων, αλλά δεν δεχόμαστε ότι θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος τρόπος να χρησιμοποιούνται μέτρα ασφαλείας και όχι να χρησιμοποιούμε τα πιο υψηλά μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι δυνατά σήμερα. Επίσης, δεν μπορεί ένα κράτο να φέρει το βάρο των ασθενειών και των προβλημάτων στον πληθυσμό λόγω του γεγονότο ότι ένα κράτο μέλο το οποίο βρίσκεται δίπλα δεν ακολουθεί αυτά τα υψηλά στάνταρτ. Ο στόχο μα είναι με αυτή την πρώτη με την οδηγία να κάνουμε ένα πρώτο βήμα προ την κατεύθυνση τη βελτίωση τη κατάσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί πολλέ προσπάθειε. Δεν πρέπει εδώ πέρα να παραμείνουμε μονάχα σε μια συζήτηση για την ε, για τι αρμοδιότητε πρέπει να δώσουμε στην Κομισιόν τη δυνατότητα να έρθει με πιο φιλόδοξες προτάσεις εν ώψη ήδη και της κατάστασης στην Ιαπωνία. Επίσης, από την Κομισιόν θα πρέπει να υπάρξει και μία μεγαλύτερη σαφήνεια και αλήθεια σε σχέση με τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με την τελική εναπόθεση των ε, αποβλήτων, κατά πόσο αυτές οι θέσεις εναπόθεσης δίνουν εγγύηση για μελλοντική ασφάλεια. Αν μετά από 50-100 χρόνια, για χρόνους οι οποίοι είναι οι χρόνοι ημιζωής των πιο ενεργών ραδιεργών προϊόντων, κατά πόσο αυτοί οι χώροι μπορούν να θεωρηθούν ασφαλείς. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιόν να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα αυτά και στην περίπτωση αυτή θα μπορούμε να έχουμε μια πιο κριτική στάση έναντι της ε, πυρηνικής ε, ενέργειας. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση όλων αυτών των προβλημάτων για να δούμε κατά πόσο θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή την ενέργεια και με ποιο τρόπο για να περιορίσουμε συγχρόνω και τις βλάβες προς την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ, λέω πρόεδρος, κύριε Ζέμπερ. Ευχαριστούμε η Επιτροπή τώρα. Έχουμε δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, την Κριστίνα Νέτσο και την κυρία Χίργεν. Δεν τους βλέπω όμως. Α, εκεί είστε. Ο κύριος Βόλφαν Χίλγερ, παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα πολυάριθμα σχόλια και τη γενικότερη υποστήριξη για την πρόταση της Επιτροπής. Το εκτιμούμε. Προηγήθηκαν εκτεταμένες βέβαια διαβουλεύσεις της πρότασης. Έχουμε συλλέξει ήδη πάρα πολλά πολύτιμα σχόλια και τα εξετάζουμε με προσοχή. Επίσης αναλύουμε με ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία, ούτως ώστε να μην υπάρξει επικάλυψη με την κείμενη ε, νομοθεσία. Κάποια από αυτά που αναφέρθηκαν σήμερα θα οδηγήσουν ακριβώς στην επικάλυψη με την ε, κείμενη νομοθεσία. Ε, για τα ορυχεία ουρανίου παραδείγματος χάρη διότι τέτοια ζητήματα ήδη καλύπτονται πλήρως από την νομοθεσία. Για την ε, ασφάλεια των χώρων τελικής διάθεσης και όλες τις υπόλοιπε δραστηριότητες και εγκαταστάσεις, η οδηγία είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Ε, ως προς την ασφάλεια, ζητείται ένα περίβλημα ασφαλείας για να καλυφθούν όλοι οι κίνδυνοι, ακόμη και όλα τα απίθανα σενάρια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια μιας δραστηριότητας ή μιας εγκατάστασης. Είναι μια εκ των... Ε, μια απαραίτητη προϋπόθεση εκ των όνου για να διατεθούν με ασφάλεια τα απόβλητα και για να υπάρχει επαρκής εποπτεία για ε, μεγάλες περιόδους. Ε, κατοχυρώνεται η ασφάλεια, καταδεικνύεται φυσικά ότι ε, κατοχυρώνεται η ασφάλεια χάρη σε αυτές τις διατάξεις και θα εμείνουμε σε αυτό το σημείο όταν να μιλάμε και για το παρελθόν στην, ε, στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων είχαμε κάποια ατυχήματα. Προτού καν οικοδομηθεί μια εγκατάσταση πρέπει να ε, τα προβλέπουμε για να ελαχιστοποιούμε ε, τους κινδύνους. Δεν μπορούμε ποτέ να αποκλείσουμε τον κίνδυνο, αλλά μπορούμε να τον ελαχιστοποιήσουμε. Επίσης, ε, χρειάζεται ε, μία διάκριση ανάμεσα στην υπέργεια αποθήκευση. Εκεί ε, υπάρχει δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης και να γίνει διάκριση λοιπόν με την παθητική ασφάλεια και την πιθανή επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Η μακροχρόνια υπέργεια αποθήκευση ενέχει κινδύνους και χρειάζεται παρακολούθηση καθώς αυξάνονται και οι επιστημονικές γνώσεις και μας επιτρέπουν να διαφυλάτουμε την ασφάλεια στην αποθήκευση. Αυτή είναι η βάση της πρότασης της Επιτροπής. Τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν εθνικά προγράμματα, εφεδρικά σχέδια για την διάθεση των αναλωμένων καυσίμων και για τη διαχείριση αυτών. Χάσαμε δύο υποθέσεις ε, ε, για τα ε, απόβλη στο δικαστήριο για τα στρατιωτικά απόβλητα. Δεν σημειώσαμε επιτυχία και είναι όντως πολύ δύσκολο το θέμα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να καλυφθούν και αυτά τα απόβλητα της αμυντικής βιομηχανίας. So uh, uh, Είπαμε και προηγουμένως ότι έγιναν ε, πολλές διαβουλεύσεις πριν καταθέσουμε την πρότασή μας και προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε τις ευέλτιστες πρακτικές ε, στην πρότασή μας. Από την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας λάβαμε δέκα συγχαρητήρια για την πρότασή μας. Δεν το περίμεναν ποτέ ότι θα είναι τόσο πλήρης η πρότασή μας. Και αυτό ισχύει και για την απαγορεύση εξαγωγών που θέλουμε να ενσωματώσουμε στην οδηγία. Είναι, έχει μεγάλη σημασία αυτό για την τελική διάθεση και σας διαβεβαιώ ότι είναι πολύ δύσκολο να υπερασπιζόμαστε αυτή τη θέση για την απαγόρευση των εξαγωγών. Σε αυτή την ε, δίνει κατάσταση που επικρατεί στην Ιαπωνία. Δεν μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε τις ιδέες σας ε, για την διαχείριση ε, των αποβλήτων ανεξάρτητα από τις αποφάσεις για το μέλλον της πυρηνικής βιομηχανίας, ε, τα υφιστάμενα απόβλητα και αυτά που παράγονται τώρα, κάποιος πρέπει να τα διαχειριστεί. Αυτή η συζήτηση για την οδηγία για τα απόβλητα θα επηρεαστεί από ε, τα ατυχή γεγονότα στην Ιαπωνία. Το σημαντικό είναι να καταδεικνύεται ότι τηρούνται οι διατάξεις ασφαλείας. Και πάλι σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και περιμένουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής σας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Χίλντε. Ο κύριος Πότς για την ε, τελική ε, παρουσίαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους για τα πολύτιμα σχόλια που έκαναν. Συμφωνώ με την κυρία Ρόσμπαχ θα πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω το θέμα της επανεπεξεργασίας των αποβλήτων και να μην θεωρούμε ότι δεν μπορώ, υπάρχει καμία πιθανή χρήση για αυτά τα απόβλητα. Ε, επίσης, ενδιαφέρον αυτό που είπε η κυρία Χάρμς, γίνονται, ε, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ε, και χαίρομαι πολύ, ελπίζω και άλλοι συνάδελφοι να βρουν χρόνο και να αφιερώσουν στο θέμα αυτό και να δεχθούν τις διαδοχικές προσκλήσεις μου για συζήτηση. Αυτή η οδηγία θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα, διότι υπάρχει μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να ρυθμίσουμε ε, ε, ενδελεχέστερα. Ή θα πρέπει να τηρήσουμε την αρχή της πρόληψης και να βρούμε απαντήσεις ε, πριν αρχίσουμε να δημιουργούμε ε, νέες ε, κατηγορίες αποβλήτων. Σίγουρα θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα και ούτως ή άλλως θα συνεχιστούν οι συζητήσεις και στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο που είναι η Α, ναι, ξέχασα λέει ο Πρόεδρος, 21η Μαρτίου 2011 είναι η καταληκτική ημερομηνία για, την, για τις τροπολογίες μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Τον Ιούνιο θα περάσει από την Ολομέλεια το σχέδιο γνωμοδότησης. Στις 12 Απριλίου θα ψηφίσουμε εδώ και στις 26 Μαΐου στην Επιτροπή Ήτρε. Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση της κυρίας Δρόσμπαχ. ΑΕΠ και πέρα από αυτό η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Παρακαλώ κυρία Ρόσμπα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ στο θέμα αυτό εν συντομία. Στην αρχή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδους εισηγητές για τον τρόπο με τον οποίο με ευέλικτο και εύκαμπτο τρόπο έχουν συνεισφέρει τις ιδέες τους για το θέμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία η οποία έχει συγκεντρώσει όλες αυτές τις ιδέες και τις έχει διατυπώσει μέσα από ένα έγγραφο εργασίας, το οποίο πιστεύω ότι μπορεί, ελπίζω ότι μπορεί να τύχει γενική υποστήριξη. Ο στόχος μας είναι να μειώσουμε τις ε, αμφιλεγόμενες και επίμαχες δηλώσεις και να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση δικτών οι οποίοι είναι μετρήσιμοι και συγκρίσιμοι. Και ελπίζω ότι θα γίνει αυτό γενικά δεκτό. Επίσης, Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτή την ε, έκθεση για το επέκεινα του ΑΕΠ με μεγάλη ταχύτητα, ώστε να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία η οποία έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή των πολιτών μας. Η ελπίδα μου επίσης είναι να υπάρξουν ενδιαφέρουσες και καινοτόμες προτάσεις και ιδέες που θα προέλθουν από την Κομισιόν μετά από την έγκριση αυτής της έκθεσης. Φυσικά τα πράγματα αυτά δεν έχουν σταθεί εύκολα. Ήταν είναι σήμερα αυτή η δεύτερη προσπάθεια που καταβάλει η Επιτροπή μας. Εγώ πιστεύω και έχω ελπίδα ότι θα γίνει κάτι γιατί υπάρχει γενική διαθεσιμότητα να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται και στην ατζέντα πολλών διεθνών οργανισμών που ζητούν να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα ως ζήτημα προτεραιότητας. Πιστεύω λοιπόν ότι τώρα κάνουμε το πρώτο βήμα προ μια κατεύθυνση που θα είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σταματήσω εδώ λοιπόν και θα ήθελα να ακούσω και τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σνέλχαρτ έχει το λόγο τώρα. Και μετά ο κύριος Πρόντι. Η κυρία Μπελιέ. Ο κύριος Σνέλχαρτ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μα είπε η συγγήτρια ότι είναι η δεύτερη προσπάθεια που καταβάλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Η πρώτη, όπως γνωρίζουμε όλοι, απέτυχε γιατί δεν υπήρχε μεγάλη ικανοποίηση ε, από τις διάφορες πολιτικές πτέρυγες στο Κοινοβούλιο. Ορισμένοι θεωρούσαν ότι ήταν ανεπαρκής η πρόταση, άλλοι θεωρούσαν ότι ήταν υπερβολικά αυτά τα οποία ζητούσαμε. Σίγουρα όμως ήταν σαφές ότι δεν, υπήρχαν, δεν υπήρχε ομοφωνία για το θέμα αυτό. Θα ήταν λοιπόν πολύ θετικά αν η συγγήτρια μέσα στα πλαίσια της νέας πρότασής της καταφέρει να εξεύρει μια πλειοψηφία η οποία θα υποστηρίξει αυτή την πρόταση και της εύχομαι κάθε επιτυχία. Τώρα, επί του πρακτέου, επί του θέματος που μας απασχολεί. Ξέρουμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό. Θέλουμε όλοι να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση για το θέμα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι η πρόταση της κυρίας Ρόσπαχ είναι απόλυτα αποδεκτή αλλά πρέπει να σας πω παράλληλα, αυτό το οποίο για μας είναι το πιο σημαντικό. Σημαντικό για μας είναι ότι το ΑΕΠ να παραμείνει στο κέντρο των δικτών που χρησιμοποιούμε. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να διευρύνουμε την έννοια του ΑΕΠ. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για αυτό. Είναι μια καλή προσπάθεια να πάμε προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν καταμετρώνται μέσα στα πλαίσια του ΑΕΠ. Αλλά εάν θεωρήσουμε το ΑΕΠ είναι η βάση της καταμέτρησης, η βάση των δικτών αυτών, θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους να καταμετρήσουμε την ε, επιρροή της ανεργίας, των ε, επιπτώσεων στο περιβάλλον και για μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Δεν θα πούμε να πετάξουμε έξω το ΑΕΠ και να ασχοληθούμε μόνο με το περιβάλλον και την ε, απασχόληση. Αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα ενσωματώσουμε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές διαφορές στον τρόπο καταμέτρησης. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια ήπια οδό μετάβασης σε νέους δείκτες, διατηρώντας πάντα στο κέντρο της ε, προσοχής μας το ΑΕΠ. Έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε την πρόταση της κυρίας Ρόσπαχ και μπορούμε να εξασφαλίσουμε και μια συμφωνία μεταξύ μας. Κάνω λοιπόν μια έκκληση προς την κυρία Ρόσπα και προς τους συναδέλφους της Επιτροπής μας να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια απόφαση η οποία θα είναι θετική και η οποία θα βελτιώσει την πρόταση της Επιτροπής ώστε να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια και μεγαλύτερη αντικειμενικότητα σε σχέση με τους δείκτες αλλά φυσικά θα πρέπει να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συνένεση για δείχτες οι οποίοι θα είναι χρήσιμοι για την Ευρώπη. Προσέξτε όμως, αν ζητήσετε πολύ γραφειοκρατικά μέτρα για την καταμέτρηση αυτών των στοιχείων, αυτό δεν ωφέλει και δεν πρόκειται να προωθήσει την έγκριση αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χώρος λέει Ο Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Ράουσμπαχ για την ε, σπουδαία εργασία της. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κλείσει σε λίγες μέρες. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σταδιακά. Με τον τρόπο αυτό ξεκινάμε μια έρευνα εις βάθος όσον αφορά την βιωσιμότητα γενικότερα. Υπάρχει μια ανάγκη για διεύρυνση της έννοιας της ε, ανάπτυξης όπου θα υπάρξει και πολιτιστική αξιολόγηση. Βέβαια αυτό παίρνει περισσότερο χρόνο. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ξεκινάμε αυτού του είδους την εμβάθυνση που είναι εξαιρετικά σημαντική. Ακριβώς επειδή μας επιτρέπει να εξετάσουμε και την ουσία της συνύπαρξής μας. Και είναι σημαντικό λοιπόν που όλα αυτά ξεκινούν εδώ στο Κοινοβούλιο, ακόμα και με τις επιφυλάξεις που υπάρχουν, αλλά μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί μια τέτοια λογική. Μια δουλειά πολύ μακρόπνοη, αλλά πιστεύω πως μπορούμε να το ξεκινήσουμε εμείς επειδή μας είναι ιδιαίτερα προσφυλής η βιωσιμότητα του πολιτισμού μας, η επιβίωση του πολιτισμού μας που περνά και από αυτή την ανάλυση. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Ρόσμπαχ για αυτή την εργασία και σίγουρα θα συμβάλλουμε όλοι. Ευχαριστώ. Dziękuję Χιτοριο Koleżanka Sandrine Bellier. Ευχαριστούμε. Η Σαντρίν Μπελιέ τώρα. Θα συμφωνεί Με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγγήτρια για αυτή τη δεύτερη απόπειρα. Βρέθη τελικά η ισορροπία νομίζω. Όχι αρκετά φιλόδοξο για τους οικολόγους, για άλλους είναι επαναστατικό ρήξη Νομίζω ότι ε, καταφέραμε, εν πάση περιπτώσει, να συμφωνήσουμε για το ότι ήδη από σήμερα και μελλοντικά θα έπρεπε να αναπτύξουμε νέα εργαλεία για να ε, μετρούμε την πρόοδο και τους διαθέσιμους πόρους. Την ανάπτυξη μάλλον και τους διαθέσιμους πόρους. Τα βασικά εργαλεία που είναι η πηξίδα μας σήμερα για την οικονομική πολιτική είναι ουσιαστικά το ΑΕΠ, και άλλα τα οποία όμως δεν είναι ικανοποιητικά, δεν επαρκούν. Διότι δεν αντανακλούν την ε, ε, πραγματικότητα στις κοινωνίες μας, τις δραγδαίες εξελίξεις, ε, δεν λαμβάνει υπόψη τις οικονομικο-περιβαλλοντικούς παράγοντες που μέσω μακροπρόθεσμα δεν συμβάλλουν στην ενίσχυση του, της πολιτιστικής ε, κληρονομιάς μας ε, και της ε, εύρωσης της οικονομικής πορείας των χωρών μας. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε σταδιακά αυτούς τους δείκτες. Δεν θα πρέπει το ΑΕΠ να θεωρείται αυτός σκοπός. Είναι ένα μεταξύ άλλων εργαλείων που θα μας επιτρέψουν να εκτιμήσουμε την ανάπτυξη τον πλούτο, τους πόρους ε, των χωρών μας, ε, που, όπου σημειώνονται, όπως σας έλεγα, ραγδαίες εξελίξεις. Θα υποστηρίξουμε αυτή την έκθεση, όπως σας έλεγα και στην αρχή. Είναι πολύ καλό σημείο κίνησης. Είναι ένα εφαλτήριο για να κάνουμε ακριβέστερες μετρήσεις, για να θεσπίσουμε, να φτιάξουμε νέα εργαλεία και θα υποστηρίξουμε την αρχική μη τροποποιημένη εκδοχή της πρότασής σας. Σας ευχαριστούμε. Η Μαρίσα Ματίας τώρα. Α, όχι, η Μαρίσα Ματίας, η Κάριν Κάντεμπεχ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που είπαν οι δύο προλαλήσαντες. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα γεγονότα της Ιαπωνίας. Βλέπουμε ότι και εκεί ο πληθυσμός βασίζεται στην ύπαρξη μιας οικονομίας. Δεν μπορούμε όμως να θεωρήσουμε ότι απλώς και μόνο η οικονομική ανάπτυξη οδηγεί σε, μια καλύτερη, σε καλύτερες συνθήκες ε, βιωτικού χαρακτήρα. Πρέπει λοιπόν όπως ελέγχθη να συνδέσουμε την ανάπτυξη με την βιωσιμότητα. Και δεν μπορεί η οικονομική ανάπτυξη από μόνη της να είναι το, το μοναδικό κριτήριο. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μια διαφορετική φιλοσοφία και αυτή πρέπει να την αναπτύξουμε και μέσα στις πολιτικές μας ομάδες. Θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι στρατηγικές μας για το μέλλον. Αν αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι μονάχα η οικονομική ανάπτυξη ή αν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα στοιχεία της αηφορίας, προστασίας του περιβάλλοντος κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε το δρόμο της βιωσιμότητας και να δούμε με ποιο τρόπο ζουν οι άνθρωποι. Ένα τέτοιο δείκτη είναι πόσα χρόνια ζει κανεί στι κοινωνίε μα σε καλή υγεία, παραδείγματο χάρη. Δεν είναι θέμα μονάχα, παραδείγματο χάρη, το να δει κανεί το προσδόκιμο επιβίωση, αλλά και την ποιότητα του προσδοκίμου αυτού και είναι πάρα πολλά γεγονότα τα οποία έχουν έρθει στο προσκήνιο με του σεισμού στην Ιαπωνία. Ευχαριστώ, η Κρίστα Κλάς. Ευχαριστώ πολύ. Να επανέλθω σε ένα ερώτημα τώρα, το οποίο ετέθη. Αυτά τα οποία έλαβαν στην Ιαπωνία ακριβώς έχουν τροποποιήσει και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής. Τώρα βλέπουμε ότι έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση στην ποιότητα ζωής από ό,τι στο παρελθόν. Εγώ χαίρομαι για το γεγονός ότι υπάρχει μια νέα προσέγγιση και υποστηρίζω και αυτό που είπε ο κύριος Σνέλχαρτ, ότι θα πρέπει στην στον πυρήνα να παραμείνει βέβαια το ΑΕΠ, αλλά φυσικά θα πρέπει να το να αυτή την έννοια για να λάβουμε υπόψη και άλλες πτυχές. Εδώ όμως υπάρχουν μια σειρά ερωτηματικών. Ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε θα πρέπει να είναι εφικτό. Και θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν. Έχει τη δυνατότητα να καταμετρήσει την ανάπτυξη με νέους δείκτες, αυτά που λέγονται στα σημεία 3, 5, 6, 7. Θα πρέπει να υπάρξουν νέοι ενδείκτες, νέα α, σταθμά και μέτρα μέτρησης, που κατά την άποψή μου δεν πρέπει να είναι άκαμπτοι δείκτες, θα πρέπει να έχουν μια ευελιξία. Θα ήθελα να ξέρω από την Κομισιόν αν, όπως ζητούμε πάντα μια έκθεση αντικτύπου, κατά πόσο θεωρεί ότι αυτά τα δεδομένα μπορούν πράγματι να καταμετρηθούν και αν μπορεί η Κομισιόν να ζητήσει λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα να τις παραδίδουν από τα κράτη-μέλη και να είναι αξιόπιστα. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο ήθελα να θέσω. Ευχαριστώ πολύ Κρίστα. Τώρα. Ο κύριος Ταταρέλα. Ναι, πολύ σύντομα. Ο κόσμος αλλάζει ταχύτατα και γι' αυτό και είναι σωστό να αλλάξουν και οι μέθοδοι μέτρησης. Ε, Συγχαρτήρια λοιπόν στην εισηγήτρια που ανέλαβε αυτήν την έκθεση. Διαπιστώνω πως ήταν δύσκολη η δουλειά γιατί είναι μια καινοτόμα έκθεση. Εύχομαι ε, γι' αυτό το θέμα η συζήτηση να συνεχιστεί εντός του Κοινοβουλίου και πέρα από την έγκριση αυτής της έκθεσης είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει όλες τις πολιτικές ομάδες και ελπίζω να υπάρξουν μάλιστα και ακροάσεις για το θέμα. Ακριβώς έτσι ώστε να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σαλβατόρε. Ήρθε η ώρα να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν, στον κύριο Τσβίλμαρ. Καλημέρα σας. Ξέρω ότι είναι η δεύτερη απόπειρα η οποία γίνεται τώρα για τα θέματα αυτά της διεύρυνσης του ΑΕΠ και η οποία από την πλευρά του Κοινοβουλίου υποστηρίζει σε γενικές γραμμές τη θέση της Κομισιόν, η ανακοίνωσή μας ήταν σαφής ότι το ΕΠ θα εξακολουθήσει να παραμένει και στο μέλλον ο πιο σημαντικός δείκτης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να διευρυνθεί και να περιλάβει πτυχές που δεν είχαν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν. Από ό,τι φαίνεται, από δημοσκοπήσεις τα δύο τρίτα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν το να υπάρξει ένα πιο ε, ευρύ έδαφος για την καταμέτρηση της ανάπτυξης. Τώρα έρχομαι στα συγκεκριμένα ερωτήματα του εφικτού και του γραφειοκρατικού άχτους. Το μόνο που μπορώ να πω εδώ πέρα, εν συντομία, είναι το εξής, ότι ακόμα και στη χρονική στιγμή κατά την οποία έγινε η ανακοίνωση της Κομισιόν, έχουμε ελέγξει τα στοιχεία για, τους, για τα κοινωνικά ζητήματα που έχουμε στη διάθεσή μας μέσω του Eurostat. Έχουμε λοιπόν τα στοιχεία από διάφορες κοινωνικές έρευνες τα οποία μπορούν να τύχουν μιας συγκέντρωσης και συμπίλησης και θα μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα για τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα της διανομής του πλούτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά οι μελέτες αυτές δεν έχουν περατωθεί ακόμα, δεν έχουν δημοσιευθεί αλλά μπορώ να σας πω ότι επί τη βάση των στοιχείων που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε καλύτερους δείκτες. Για το περιβάλλον τώρα, χρησιμοποιούμε, εργαζόμαστε για τον περίφημο συνθετικό δείκτη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, αλλά η κατάσταση των δεδομένων δεν βρίσκεται στο επίπεδο που εμείς θα θέλαμε να έχουμε. Ακόμα θα πρέπει να βρούμε πιο καινοτόμου τρόπους για μια καλύτερη συλλογή δεδομένων σε σχέση με το περιβάλλον. Τίθεται, όπως ελέγχθη, και το θέμα της γραφειοκρατίας και του γραφειοκρατικού άχθους. Εδώ θα πρέπει να έχουμε ίσως μια διαφορετική προσέγγιση. Όλο και περισσότερο έχουμε στατιστικές από επίσημες αρχές, αλλά και από άλλες πηγές, και όλο και περισσότερο θεωρούμε ότι αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία για λήψη αποφάσεων, για εκθέσεις αντικτύπου παραδείγματος χάρη. Όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται από το γεγονός ότι τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά στοιχεία συλλέγονται σε παράλληλο επίπεδο και συγχρόνως και είναι αρκετά αξιόπιστα για να επιτρέψουν την λήψη αποφάσεων. Πρέπει λοιπόν να δούμε τη συλλογή αυτών των στατιστικών στοιχείων ως μια απαραίτητη επένδυση για την καλύτερη προετοιμασία των αποφάσεων και όχι απλώς σαν μια πρόσθετη επιβάρυνση ή μια πρόσθετη γραφειοκρατία η οποία έχει μόνο εχει μοναδικο χαρακτηρα Ευχαριστώ. Ο Χώρστα Σνέρχαρτ. Ένα ακόμα ερώτημα θέλω να θέσω στην Κομισιόν. Γιατί με απασχολεί αυτό το θέμα και συμφωνώ με αυτό που λέτε. Μιλάτε για μια καλύτερη κατανομή ε, εισοδήματος, παραδείγματος χάρη. Πώς βλέπετε το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς θα μπορούσε να υπάρχει μια κοινή ρύθμιση, παραδείγματος χάρη, που θα λαμβάνει υπόψη την κατανομή εισοδήματος. Σας ευχαριστώ, λέει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δει διασαφηνίσω περισσότερα τα πράγματα για το πώς η Κομισιόν θέλει να προχωρήσει να αντιμετωπίσει το θέμα της κατανομής εισοδήματος. Απλώς μας απασχολεί πώς κυμαίνονται συνθήκες ζωής σε διάφορα στρώματα του πληθυσμού και το ερώτημα του πώς αυτό μπορεί να τροποποιηθεί εν καιρό αυτό θα έχει νόημα μονάχα όταν έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Δηλαδή πρέπει πρώτα να έχουν συλλεγεί οι πληροφορίες προτού υπάρξει μια διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης κατανομής εισοδήματος, το οποίο φυσικά είναι μια πολιτική απόφαση σε τελική ανάλυση. Σας ευχαριστώ. Στρέφομαι προς την εισηγήτρια. Θα θέλατε να πάρετε το λόγο, κυρία Ρόσμπαχ. Παρακαλώ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, θα ήθελα να κάνω ένα τελικό σχόλιο. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσους παρενέβησαν για την επικοδομητική του στάση. Και κύριε Σινέλχαρτ, όχι, Δεν σκέφτηκα ποτέ την κατάργηση του, GDP, του ΑΕΠ, συγγνώμη, την αντικατάστασή του με κάτι άλλο. Όχι. Απλώς ε, θα ήθελα να χρησιμοποιηθούν και νέοι δείκτες, όπως για παράδειγμα όταν πρόκειται για την ενέργεια. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο μία μονάδα μέτρησης. όπως για την ενέργεια δεν μπορούμε να επιβιώσουμε μόνο με το πετρέλαιο, πρέπει να διαφοροποιηθούμε. Και περί αυτού πρόκειται και εδώ. Η προσέγγιση σκοπεύει, θέλει μάλλον να συμπεριληφθούν στις μετρήσεις όσο γίνεται περισσότερες πτυχές. Και δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε σε κάποιο οριστικό αποτέλεσμα, διότι όπως ήδη υπόθηκε ο κόσμος διαρκώς αλλάζει και γι' αυτό και οι μετρήσεις αυτές θα αλλάζουν συνέχεια. Και οι μονάδες μέτρησης θα πρέπει να ανανεώνονται διαρκώς. Βλέπω ωστόσο ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, ε, όχι μόνο εδώ για την Ευρώπη, αλλά εμείς εστιάζουμε την προσοχή μας στην Ευρώπη, αλλά είναι ένα θέμα επί το οποίο θα συνεργαστούμε στενά με την Κομισιόν. Νομίζω πως είναι ένας τομέας στον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες για να φτάσουμε σε αποτελέσματα που θα ωφελήσουν ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι λοιπόν πολύ θετική αυτή η ατμόσφαιρα και συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους του Κοινοβουλίου ότι όντως θα πρέπει να μπορέσουμε να εμπλέξουμε και την κοινωνία και να κάνουμε και κάποιες ακροάσεις εδώ στο Κοινοβούλιο για να δούμε πού οδεύουμε ως κοινωνία, τι προσαρμογές θα πρέπει να κάνουμε καθώς προχωράμε. Προσβλέπω λοιπόν σε μια συζήτηση, προσβλέπω στη βοήθειά σας ώστε το έγγραφο αυτό να αποτελέσει ένα καλό σημείο εκκίνησης για πολλές στιγμές που θα περάσουμε μαζί στο μέλλον για αυτό το σπουδαίο θέμα. Ευχαριστώ κυρία ε, Ρόσμπαχ. Κλείνει η συζήτηση για αυτό το θέμα και το επόμενο σημείο, α, πριν περάσω στο επόμενο σημείο, να σας πω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 21η Μαρτίου 2011 στις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε εδώ στις 19 Απριλίου και στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Επόμενο σημείο είναι το 27. Ανταλλαγή απόψεων με την εκπρόσωπο της Επιτροπής για την παρουσία χαμηλών ποσοτήτων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο τρόφιμα. Να δώσω το λόγο στην Επιτροπή Έχουμε τον διευθυντή Έρικ Κούδελε. Εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η γενική μας διευθύντρια, η κυρία Τεστόρη Κότζη, έπρεπε να είναι εδώ κανονικά, αλλά είχαμε συμβουλαλλαγή για την κλωνοποίηση όλο το βράδυ και προεδρεύει ε, σε μια διάσκεψη για του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού που συνδιοργανώνουμε με το Κοινοβούλιο, γι' αυτό και δεν παρίσταται στη συνεδρίασή σας. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιβάλλοντος, πάντως μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτή την πρόταση που ψηφίστηκε με ειδική πλειοψηφία στη Μόνιμη Επιτροπή για τη Διατροφική Αλυσίδα στις 22 Φεβρουαρίου και άρα κατατίθεται τώρα στο Κοινοβούλιο στα πλαίσια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Ε, έχετε τρεις μήνες για να γνωμοδοτήσετε βάσει της διαδικασίας. Ε, μηδενική ενοχή είχαμε στο παρελθόν ε, για τις εισαγωγές γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που δεν έχουν αποτελέσει το αντικείμενο απόφαση ε, έγκριση ε, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. μηδενική ανοχή δημιουργούσε διάφορα προβλήματα διότι τα κράτη-μέλη δεν είχαν ε, ίδιες μεθόδους διάγνωσης αυτό δημιούργησε διάφορες αβεβαιότητες ε, για τους εμπορικούς, τους οικονομικούς φορείς. Ε, ήταν μια αρχή ε, ευεφάρμοστη, αλλά παρουσίαζε δυσκολίες ως προς τεχνική υλοποίησή της, διότι γενετικά τροπημένοι οργανισμοί μάλλον δημητριακά με τέτοιους ε, απαγορευμένους ε, οργανισμούς αναλύονταν στους μεθοριακούς σταθμούς και έφευγαν ολόκληρα σκάφη φορτωμένα προς την χώρα προέλευσης. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε λοιπόν μια πρόταση που εξετάζεται τώρα με στόχο την εναρμόνιση των ελέγχων στην εισαγωγή κυρίως. προβλέπει η απόφαση αυτή μια σειρά πρωτοκόλων για τη δειγματοληψία, για τις δοκιμές με διάφορες διαγνωστικές μεθόδους. Τα βλέπετε στο παράρτημα, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Le plus petit Προσδιορίζει λοιπόν το ελάχιστο επίπεδο γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που μπορεί να εντοπιστεί βάσει της μεθόδου που προβλέπεται, μιας αξιόπιστης, αξιόπιστης ε, ε, μεθόδου που ε, δεν μπορούν να αμφισβητήσουν οι εξαγωγές της Βορείου ή Νοτιού Αμερικής. Αυτό είναι σημαντικό, διότι στο παρελθόν όταν ε, ένα κράτος μέλος, ένα φορτίο δημητριακών είχε θετικό αποτέλεσμα που προσέγγιζε το επίπεδο της μηδενικής ανοχής, ε, γινόντουσαν, ε, ε, υπήρχαν ατέρμονες αντεγκλήσεις, αν θέλετε, ανάμεσα στους ειδικού ε, του, των δύο κρατών, της εισαγωγής και της εξαγωγής, δηλαδή των εμπορευμάτων. Τώρα θέσαμε το όριο στο 0,1% ε, για την ανοχή αυτών των οργανισμών. Έτσι παρέχονται όλα τα ηχέγγυα, είναι αξιόπιστη μέθοδος, αξιόπιστα μπορούμε να εντοπίσουμε αυτούς τους οργανισμούς. Είναι το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε με την βέλτιστη τεχνική που προβλέπεται στο παράρτημα. Αυτή η τεχνική έχει κυρωθεί από το εργαστήριο αναφοράς της Ένωσης για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς είναι ε, ε, η πιο ευαίσθητη, ακριβής μάλλον μέθοδος. Και όταν έχει εντοπιστεί αυτό το ελάχιστο ποσοστό δεν υπάρχει περιθώριο αμφισβήτησης από κάποιον τρίτον. Συνοδεύεται από τρεις όρους δε η πρότασή μας. Πρώτον, ο οργανισμός θα πρέπει να έχει εγκριθεί στην τρίτη χώρα που εξάγει προς την Ένωση. Άρα ε, έχει γίνει επιστημονική αξιολόγηση σε αυτή την τρίτη χώρα. Δεύτερος όρος ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση από την ε, υπηρεσία μας για την ασφάλεια των τροφίμων, από την ΕΦΣΑ δηλαδή. Γίνεται μια σειρά αξιολογήσεων και δοκιμών από πλευράς ε, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων ή έχει πάρει στο παρελθόν έγκριση ε, ο συγκεκριμένος οργανισμός, αλλά έχει εκπνεύσει η έγκριση. Τρίτος όρος, η ΕΦΣΑ θα πρέπει να μας πει ότι τα υπολείμματα αυτά, ε, ε, κάτω του 0,1% πρέπει να αποδείξουν ότι δεν συνιστά αυτό κίνδυνο για τους ανθρώπους, για τα ζώα ή για το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντική η όρη αυτή. Δεν δίνουμε μια λευκή επιταγή για όλους τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που μπορεί να υπάρχουν από τον κόσμο. Είναι αυστηρά προσδιορισμένη αυτή η όρη και ούτως ή άλλως συνεχίζονται και αξιολογήσεις από την Ευρωπαϊκή ε, Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγουμε 33 εκατομμύρια τόνους σόγιας του χρόνου κατά μέσο όρο, και 4 εκατομμύρια τόνους καλαμπόκι, κυρίως από την Αργεντινή, από τη Βραζιλία και από τη ΣΥΠΑ. Το μεγαλύτερο, μάλλον σχεδόν ολόκληρες αυτές οι ποσότητες, προορίζονται για ε, ζωοτροφές. Ένα μικρό κομμάτι χρησιμοποιείται για ε, την διατροφή των ανθρώπων, ε, κυρίως ο αραβόσιτος, αλλά ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι αυτών των ε, ποσοτήτων προορίζεται για τους ανθρώπους. Ο στόχος της πρότασης αυτής είναι η εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρειάζονται κυρίως ε, τον αραβόστο και τη σόγια για τις ζωοτροφές, στα, στις μονάδες εκτροφής, τα πουλερικά, η χείρη, τα βοηδή κυρίως. Οι εισαγωγείς λοιπόν αυτοί να έχουν στη διάθεσή τους ένα σαφές ακριβές ε, νομικό πλαίσιο, ώστε ε, με τους συναδέλφους τους από τις τρίτες χώρες, τους εξαγωγείς, να μπορέσουν να λειτουργούν βάσει αυτού του τεχνικού πλαισίου, τόσο ώστε να μην φτάνουν τα φορτία με τα σκάφη στα σύνορα και να επιστρέφουν πίσω όταν είναι θετική η διάγνωση. Αυτό το 0,1% το αναλυτικό μηδέν, έτσι ονομάζεται αυτό, δηλαδή είναι το ελάχιστο ποσοστό στο οποίο μπορούμε να φτάσουμε με κάποια διαγνωστική μέθοδος, ε, το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κάποιον ε, ε, ειδήμονο. χάρη στη μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό του ποσοστού. Η επιτροπή σας είπε ότι ψήφισε την πρόταση στις 22 Φεβρουαρίου και στις 14 ε, Μαρτίου διαβιβάστηκε η πρόταση στο Κοινοβούλιο και το ε, ε, Συμβούλιο ούτως ώστε εντό τριών μηνών, όπως προβλέπετε από την διαδικασία, να γνωμοδοτήσετε και εσείς. πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά. Και τώρα μπορούμε να συζητήσουμε. Est-ce qu'il y a des questions au représentant de, de la Commission Έχετε ερωτήσεις στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Όχι. Όλα είναι ξεκάθαρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Le, le date, la date pour donner des η ημερομηνία για να εκφράσετε αντιρρήσει είναι στις 30, η 30 Μαρτίου το μεσημέρι στις 12. Merci, euh, euh, monsieur, Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουντελέ. Επόμενο σημείο στην ημερήσια μας διάταξη είναι η συζήτηση για την κοινή γεωργική πολιτική στον ορίζοντα του 2020. Απάντηση στις προκλήσεις του μέλλοντος καθώς και τις μελλοντικέ ανάγκες στον τομέα των φυσικών πόρων. Η συγγήτρια μας είναι η κυρία Κάντενμπακ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ja, herzlichen Dank. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η απαρχή αυτής της ε, συζήτησης είναι η συζήτηση για την τροποποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής μέσα σε ένα διαφορετικό παγκόσμιο πλαίσιο όπου έχει παγκοσμιοποιηθεί πολύ περισσότερο η παραγωγή τροφίμων και όπου έχουμε νέες αναδυόμενες χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα και που φυσικά όλα αυτά επηρεάζουν και την ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική. Έχουμε ζητήσει συζητήσει πάρα πολλέ φορέ για τι βιολογικέ προοπτικέ σε σχέση με τη γεωργία, τα προβλήματα διάβρωση του εδάφου κτλ. Ο στόχο μα είναι να αντιμετωπίσουμε θέσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τη σύνδεση του, της γεωργικής παραγωγής με το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Και φυσικά δεν πρόκειται να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος. Ο στόχος μου στην έκθεση αυτή είναι να καλύψω όλες τις πτυχές που είναι σημαντικές για την Επιτροπή περιβάλλοντο. Περιβάλλοντος. Έχουμε ένα περιορισμένο αριθμό λέξεων για τις γνωμοδοτήσεις μας και είναι φανερό ότι εγώ δεν μπορώ να καλύψω όλα αυτά τα, στοιχεία. Εγώ θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την άποψη των συναδέλφων και είμαι απόλυτα ανοιχτή σε περαιτέρω συζητήσει για να μπορέσω να εμβαθύνω ακόμα περισσότερο σε ορισμένα θέματα. Αυτά τα οποία εγώ έχω παρουσιάσει στα πρώτα σημεία της γνωμοδότησής μου είναι ότι πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε τους στόχους της ε, διατροφής του πληθυσμού με αηφόρες πολιτικές γεωργίες, το ότι είναι αηφόρο, είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά στην Επιτροπή μας σε σχέση με τη γεωργία και επίσης παράλληλα πρέπει να υπάρξουν νέες μορφές εξοικονόμησης ενέργειας οι οποίες θα ακολουθηθούν με τρόπο ή θελημένο και επίσης να υπάρξει και περιορισμός της χρήσης χημικών λιπασμάτων. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει το οικοσύστημά μας για να τις χρησιμοποιήσουμε με τρόπο αποτελεσματικό χωρίς να δημιουργούμε κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και συγχρόνως να κάνουμε την προσπάθεια να εξασφαλίσουμε και την διατήρηση της βιοπικιλότητας. Θέλουμε να στραφούμε κατά της εξάντησης των φυσικών πόρων και τη διάβρωσης και υποβάθμισης τη ποιότητα των αρρωσίμων εδαφών. Επίσης με το πρόγραμμα έρευνας της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης βρίσκουμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν περισσότερο, να υπάρξει περισσότερη έρευνα ώστε να μειωθεί και η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2025. Οι γεωργοί μας πρέπει και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να έχουν παραγωγή φτηνότερων τροφίμων για τον πληθυσμό, αλλά θα πρέπει να προστατεύσουν και το περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι αυτή η πλευρά έχει ιδιαίτερο, ιδιαίτερη σημασία για μας, γιατί εξάλλου έχει αλλάξει και η γεωργία σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι δεδομένο ότι ο γεωργός μονάχα πρέπει να παράγει, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσει και για τη δική του διάρκεια ζωής αλλά και για τις επερχόμενες γενναίες να διατηρήσει την ποιότητα των εδαφών και όχι μονάχα να περιοριστεί στην ε, βραχυπρόθεσμη κερδοφορία. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και στα πλαίσια τη τρέχουσα μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη και ασφάλεια για την γεωργία. Αυτό όμω σημαίνει και μεγαλύτερη ασφάλεια για τι θέσει εργασία στη γεωργία. Ο Επίτροπο κ. Τσόλο έχει ανακοινώσει ότι αυτοί οι οποίοι εργάζονται για την προστασία της φύσης θα πρέπει να έχουν και μεγαλύτερη αμοιβή για την εργασία τους από αυτούς οι οποίοι δεν προστατεύουν την φύση. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια μεγαλύτερη έμφαση στη λεγόμενη διασταυρούμενη συμμόρφωση και να υπάρξει και μια μεγαλύτερη ε, απόδοση πριν σε αυτούς οι οποίοι προστατεύουν περισσότερο το περιβάλλον. Ένα στοιχείο το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην γνωμοδότησή μου είναι και το θέμα της βιοπικιλότητας. Εδώ πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση. Αντιμετώπιση λοιπόν της βιοπικιλότητας και των κινδύνων που προκύπτουν για αυτήν από την κλιματική αλλαγή και όπως είπε και η Κοψιόν έχουμε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στην Ευρώπη που υποστηρίζει μια τέτοια προσέγγιση, επομένως βρισκόμαστε σε έδαφος ασφαλές, θα πρέπει να περιορίσουμε για αυτό το λόγο την ε, χρησιμοποίηση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, κάτι το οποίο το επιθυμεί και η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού στην Ευρώπη. Ζητούμε λοιπόν από την Κομισιόν να σκεφτεί καλύτερα ποιες είναι οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν για να υπάρξει η μικρότερη δυνατή χρήση μη κυβερνητικών, μη, συγγνώμη, μη, ε, η μικρότερη δυνατή χρήση γενικά τροποποιημένων οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ευχαριστώ. Mm. Σας ευχαριστούμε κυρία Κάντενμπαχ. Η Σαντρίν Μπελίε τώρα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Κάντεμπαχ για το σχέδιο έκθεσης. Σας ευχαριστούμε. Επιθυμείτε να έχει ορίζοντα το 2020 η κοινή γεωρική πολιτική, να έχει ανθρώπινο πρόσωπο και να προστατεύει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Συγχαρητήρια για τις τρεις εναλλακτικέ λύσει ε, της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2010 σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής θα λέγαμε τα εξής. Οι οικολόγοι μπορούν να δεχτούν μόνο την δεύτερη εναλλακτική λύση και χαιρόμαστε, δεν το κρύβω, που η συγγήτρια, η κυρία Κάντενμπαχ, συμφωνεί μαζί μας ή τουλάχιστον αυτό προκύπτει από το σχέδιο έκθεσης. Παρ' όλα αυτά, οι οικολόγοι το είπατε κι εσείς, θεωρούν ότι δεν είναι πλήρης η έκθεση. Είναι ατελής και θέλουμε να επανεισάγεται κάποια σημεία, διότι κρίνουμε ότι είναι καθοριστική σημασία. Πέντε είναι αυτά. Πέντε σημεία πρέπει να επανεισάγεται. Υπάρχει ένα σημείο επίσης όπου διαφωνούμε και τέλος... Εκ μέρους της κυρίας Χάση που δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα, να σας υποβάλλω και ε, μία τροπολογία. Τι θέλουμε να επανεισάγουμε με στην έκθεση. Πρώτον, οι μικρές μονάδες θα πρέπει να έχουν μία απλή και βελτιωμένη στήριξη για την ανταγωνιστικότητά τους και τη βιωσιμότητα της υπαίθρου, να μειωθεί το διοικητικό άχθος και να προαχθούν οι πρακτικές που νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, σέβονται περισσότερο το περιβάλλον σε σχέση με τις μεθόδους ε, εντατικής καλλιέργειας. Ε, κατόπιν, μέσα στην έκθεση θα θέλαμε να τονίσουμε ότι υποστηρίζουμε τη χρηματοδότηση μιας νέας κοινή γεωργικής πολιτικής που θα βασίζεται σε ένα μοντέλο που συμπεριλαμβάνει τις πληρωμές για ε, τη βιολογική καλλιέργεια, για την καλλιέργεια υψηλής προστιθέμενης αξίας ε, ή για την καλλιέργεια ε, υπό ειδικού όρους στις περιοχές προστατεύονται από την οδηγία Natura. Οι εντατικές ε, καλλιεργητικές μέθοδοι επηρεάζουν την υγεία των ζώων, τη διατροφική ασφάλεια και το περιβάλλον και έτσι θέλουμε η κοινή γεωργική πολιτική να ταχθεί υπέρ πρακτικών που σέβονται το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Θέλουμε με σαφήνεια να τονιστεί αυτό μέσα στην έκθεση. Επίσης, θα θέλαμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε σχέση με τη σημασία που έχει το μέλλον της βιολογικής ε, καλλιέργειας. Και τέλος, η σημασία της βιοποικιλότητας, η βιοποικιλότητα για τις καλλιέργειες, για τις ποικιλίε που καλλιεργούνται ε, και για την πανίδα έχουν ιδιαίτερη σημασία και όταν μιλάμε για την βιοποικιλότητα αυτό που διακυβεύεται είναι ο πλούτος που έχουμε από τις φυτικές ποικιλίε ε, και τα ζωικά είδη. Ε, les écologistes aujourd'hui η οικολόγια σήμερα δεν θέλουν να συμπεριληφθεί η γεωργία στις αγορές, στα χρηματιστήρια του άνθρακα. Μας δημιουργεί πρόβλημα αυτό. Ε, θα θέλαμε σήμερα να επιβληθεί ένα σύστημα που να μην να αποθαρρύνει την ε, κερδοσκοπία, την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία στα χρηματιστήρια αυτά des marchés dans le marché ο κίνδυνο να ενισχυθεί περαιτέρω η κερδοσκοπία για τα διατροφικά είδη. Όπως σας έλεγα, εμεί ανέκαθεν εντασσόμαστε. Σε αυτό δεν το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία. Όπως και η συνάδελφος Χάση, θα θέλαμε μέσα στην έκθεση να αναφερθούμε στο πρόβλημα της καλλιεργίας ε, της γεωργίας ε, στη Βαλτική θάλασσα. Είναι από τις ε, πιο μολυσμένες θάλασσες του κόσμου η Βαλτική θάλασσα. Θα υποβάλουμε τροπολογίες για όλα αυτά τα σημεία από την πολιτική μας ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπελιέ. Και το λόγο έχει η κυρία Αντωνέσκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε απόλυτη επίγνωση κύριε Πρόεδρε του δυναμικού της γεωργίας στην Ευρώπη αλλά και του ζωτικού ρόλου που έχει για την επίτευξη των στόχων του περιβάλλοντος και για τη δημιουργία δημοσίων αγαθών και επίσης για τη διατήρηση της δημόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό συγχρόνως. Όταν μιλάμε για τη γεωργία και για το μέλλον της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δώσουμε έμφαση στην καινοτομία και την απλοποίηση. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο τη ζωή των γεωργών με το να τους θέτουμε πρόσθετο διοικητικό ε, και γραφειοκρατικό άχθος αρκετά προβλήματα έχουν. Θέλουμε να υπάρξει μια πιο απλοποιημένη και πιο ισοδίκαια πολιτική. Θέλουμε να βρούμε λοιπόν μια σωστή ισορροπία μεταξύ των στόχων που θέλουμε να επιτύχουμε και του διοικητικού βάρους που θα πρόκειται. Πρέπει να έχουμε ασφαλή τρόφιμα, πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον, πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία και την ευμάρεια των γεωργών και την εδραίωση της τοπικής οικονομίας. Και ο στόχος μας είναι να έχουμε προϊόντα ε, γεωργικά τα οποία έχουν υψηλή διατροφική αξία και υψηλή ποιότητα. Γι' αυτό το λόγο η αντιμετώπιση της γεωργίας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει ζητήματα τα οποία θα έχουν μονάχα τεχνοκρατικές και τεχνολογικές λύσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πτυχές της ανθρώπινης κατανάλωσης και την πολύπλοκη αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητος και της ανθρώπινης υγείας. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω, θα παρουσιάσουμε και τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Κρίστα Κλάς έχει και το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέροντα στόχο το οποίο έχει θέσει η κυρία Κάδεμπαχ και αξίζει τον κόπο να σκεφτούμε πολύ περισσότερο για τα θέματα αυτά. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ξεχνάμε πάρα πολύ. Έχουμε μια κοινή αγροτική πολιτική η οποία στην αρχή ήταν η απαρχή και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε κοινότητα. Έχει περάσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις η κοινή αγροτική πολιτική, ώστε, όπως είπε και η κυρία Αντωνέσκου, να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και το ρόλο των γεωργών. Οι γεωργοί δεν παράγουν μονάχα προϊόντα, αλλά ο στόχος τους είναι να δώσουν στην Ευρώπη υγιή προϊόντα και όχι μονάχα τροφιμικά προϊόντα πρέπει να εξασφαλίσουν όχι μόνο την παραγωγή τροφίμων, αλλά και το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό πλαίσιο της γεωργίας στην Ευρώπη και αυτά δεν πρέπει να τα παραγνωρίζουμε. Όλο αυτό το συνολικό οικοδόμημα έχει δημιουργηθεί σταδιακά με τα χρόνια στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής, γεωργικής πολιτικής και έχουμε υποστηρίξει την γεωργία και οικονομικά παρά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί ε, μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα οι επιδοτήσεις προς τη γεωργία. Αυτή τη στιγμή παίζει ένα προεξάρχοντα ρόλο σε όλα αυτά το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, του πολιτιστικού πλαισίου, της διατήρησης θέσεων απασχόλησης και η παραγωγή υγιεών, υγιών τροφίμων. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πια τόσο υψηλή η χρηματοδότηση της γεωργίας. Πιστεύω όμως ότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουμε την ε, υγεία των ε, τροφίμων τα οποία ε, παράγονται και την σημασία του να διατηρηθεί άμομο το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται η παραγωγή αυτών των τροφίμων και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε και ποια θα είναι τα μελλοντικά βήματα για την γεωργία και το αγροτικό πανόραμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να έχουμε όλο και περισσότερους κανονισμούς. Ειδικά οι γεωργοί <clears throat> έχουν πάρα πολλές προδιαγραφές οι οποίες τους περιορίζουν για την παραγωγή των τροφίμων τα οποία θα πρέπει να είναι <clears throat> πιο η Ευρώπη θέλει να εξασφαλίσει λοιπόν την υγεία των καταναλωτών και την ε, προστασία του περιβάλλοντος και αυτό είναι το στοιχείο στο οποίο εμείς πρέπει να εστιάσουμε πολύ περισσότερο ως Επιτροπή Περιβάλλοντος. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα καθήκοντα των ε, γεωργών τα οποία μέσα στα πλαίσια της διασταυρούμενης συμμόρφωσης πρέπει να τα τηρήσουν. Το ξέρουν όλοι τι θα πει cross compliance στη Γερμανία, ακόμα και δεν ξέρουν άλλες γλώσσες. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι αυτά τα καθήκοντα ισχύουν σε όλα τα κρατήρια της ε, χώρας μου και σε όλες τις χώρες. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σκεφτεί η Κομισιόν αν θα πρέπει να βρει κάποιο τρόπο να ασκείτε μια πιο γενική εποπτεία για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται η, λαμβάνει η χώρα η διασταυρούμενη συμμόρφωση στα κράτη-μέλη, γιατί βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχουν μεγάλες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται αυτός ο κανόνας της διασταυρούμενης ε, συμμόρφωσης. Θα πρέπει η Κομισιό λοιπόν να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ένα ισόπεδο γήπεδο, ότι εφαρμόζεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι ισόμορφος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης μας ενδιαφέρει η λεγόμενη ε, ολοκληρωμένη γεωργική δραστηριότητα, αυτό σημαίνει και προστασία φυτοϊγειονομική. Όταν μπαίνουμε λοιπόν στο γενικό αυτό χώρο της ε, βιοπικιλότητος και της προστασίας των γεωργικών προϊόντων, θα πρέπει και εκεί να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει η απαραίτητη αντιμετώπιση και στην, στον δεύτερο πυλώνα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Το έβδομο σημείο που αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και την ε, συμπερίληψη των προσπαθειών της, Γερμα... Γεωργίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εδώ είναι κάπως δύσκολο αυτό, διότι δεν έχουμε ακόμα μετρήσιμα στοιχεία τα οποία μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό δεν είναι κάτι λοιπόν το οποίο εγώ μπορώ να υποστηρίξω. Το ίδιο ισχύει για το σημείο 9. Ήδη έχουμε μιλήσει με την Κομισιόν για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Νομίζω ότι δεν έχει εξαντληθεί ακόμα η συζήτηση με την Κομισιόν. Θα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση σε επίπεδο εμπεριστατωμένο και όχι απλώς να πούμε ότι απορρίπτουμε τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς συλλήβδιν. Θα ήταν καλύτερο να έχουμε μια ευρύτερη συζήτηση με την Κομισιόν αλλά σε μια άλλη ε, επιτροπή σε ένα άλλο χώρο Πρέπει φυσικά να συζητήσουμε και την πρόταση του Επιτρόπου Τσόλος να έχουμε μια καλύτερη σύνδεση με την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραγνωρίσουμε αυτά που προσφέρουν οι γεωργοί μας σήμερα και είναι σημαντικό να δώσουμε έμφαση καταρχήν σε αυτά τα οποία έχουμε τώρα, στο να υπάρχει σωστός έλεγχός τους και να ε, έχουμε έτσι από την πλευρά της Επιτροπής Περιβάλλοντος μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Κλάς, δύο ακόμα ομιλητές. Ο Chris Davis. Ο Σας ευχαριστώ. Θα κάνω δικά μου σχόλια και έχω σχόλια συναδέλφου που δεν μπορεί να είναι παρόν. Να ευχαριστήσω την κυρία Γκάντεμπαχ για την ε, εργασία της, για το ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι θα έχουμε ασφάλεια ε, τροφίμων αλλά και ασφαλή τρόφιμα αλλά και την ε, διάσταση την αγροτική πώς προστατεύουμε την αγιοργική ζωή πώς ε, εξασφαλίζουμε ότι προστατεύουμε και αυξάνουμε την βιοποικιλότητα και επίση υπάρχουν και θέματα ευρύτερα από την Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποφύγουμε το γεγονό ότι η δική μα πολιτική επηρεάζει τι τιμέ των τροφίμων σε ολόκληρο τον κόσμο και τη σχέση μα με τι στοχότερες χώρε. Εφόσον εξετάζουμε την κοινή γεωργική πολιτική, μήπω πρέπει να θυμηθούμε και πόση γραφειοκρατία απαιτούμε από του γεωργού, έτσι ώστε αυτοί να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα που δίνουμε. Δεν πρέπει αυτό να το ξεχνάμε. Έχουμε επίσης ε, πολύ καλά παραδείγματα στην Ευρώπη υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, αλλά και ταυτόχρονα πολύ κακικών προδιαγραφών. Πώς μπορούμε λοιπόν να μάθουμε από τις καλύτερες πρακτικές. Ε, δεν θα πρέπει να δεσμεύσουμε τους γενικά τροποποιημένους οργανισμούς μόνο εδώ. Θα πρέπει να ε, τους εξετάσουμε σε, άλλο, σε άλλη έκθεση. Δεν θα υποστηρίξουμε λοιπόν την παράγραφο 9, αλλά θα σίγουρα θα υποστηρίξουμε την 10 που μιλά για έρευνα, για καινοτόμους τρόπους καλλιέργειας της γης, ε, μεγάλο δυναμικό για το μέλλον. Και τώρα ε, κάποια σχόλια δικά μου, το θέμα των επιδοτήσεων και του κατά πόσο θα πρέπει να πληρώνουμε στην κοινή γεωργική πολιτική με τον τρόπο που κάνουμε μέχρι σήμερα. Συχνά ε, έχει υποστηριχθεί ως ένα μέσο προστασίας των μικρών οικογενειακών αγροκτημάτων, ιδιαίτερα στη Γαλλία. Οι Γάλλοι έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το επιχείρημα. Αλλά εγώ εξέτασα τι συμβαίνει και δεν είναι επιτυχές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο εγώ δούλευα σαν φοιτητή σε ένα αγρόκτημα, σε ένα αρρώσιμο κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου και πέντε πλήρως απασχολούμενοι διαχειρίζονταν 200 ε, εκτάρια. Τώρα έχουν κλείσει ένα σωρό αγροκτήματα. Τώρα ένα αγρόκτημα είναι χίλια εκτάρια με τρεις ανθρώπους μόνο. Φαντάζομαι το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία οι τα οικογενειακά αγροκτήματα έχουν περιοριστεί και τα περισσότερα χρήματα πάνω στους μεγάλους βαρώνους γύρω από το Παρίσι. Άντε και καμιά 200 χιλιόμετρα πιο πέρα. Άμεσες πληρωμές ή επιδοτήσεις στα αγροκτήματα, ωστόσο στην ουσία τι κάνουμε, ε, υποσκάπτουμε την ελεύθερη αγορά οι τιμέ των τροφίμων είναι ήδη πολύ ψηλέ και θα μείνουν ψηλέ. Αν σταματήσουμε να επιδοτούμε, οι τιμέ των τροφίμων θα εξισορροπηθούν. Δεν πρέπει να βάζουμε χρήματα σε μη βιώσιμε δραστηριότητε να αφήσουμε την αγορά να καταλήξει στο δικό της ε, επίπεδο. Αλλά αυτό διχάζει σίγουρα την ομάδα μου και θα διχάσει και το Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ πολύ πάντω για την έκθεση. Dewisowi. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντέιβις. Ο κύριος ε, Ρώση. Σας ευχαριστώ πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο για να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί ε, κάνει διάφορα ενδιαφέροντα σχόλια. Θέλω όμως να ζητήσω ότι από την ε, εισηγήτρια να είναι λίγο πιο ε, σαφής και απαιτητική. Να ζητήσουμε, για παράδειγμα, ε, την εγγύηση αυτών των ε, αγροκτημάτων που για μας είναι σημαντικά. Αυτά τα αγροκτήματα, τα ποιοτικά, τα ορεινά αγροκτήματα, αυτά που προστατεύουν το περιβάλλον και προσπαθούν να περιορίσουν την ρήπανση. Να ζητάμε λοιπόν να παραμείνει τουλάχιστον ένα προπολογισμό ίδιο με τον προηγούμενο, γιατί μέγας κίνδυνο είναι ότι θα μειωθεί το κονδύλι. Γιατί σε σχέση με την προηγούμενη κοινή γεωργική πολιτική έχουμε αυξηθεί από 15 σε 27 χώρε. Ήδη δηλαδή θα περιοριστούν τα κονδύλια. Εάν δεν καταφέρουμε να διατηρήσουμε και τον κατάλληλο επίπεδο στον προπολογισμό, κινδυνεύουμε να ματαιώσουμε κάθε απόπειρα να βελτιώσουμε το ε, την ποιότητα της γεωργίας. Ζητάμε δηλαδή δέσμευση από τη μια πλευρά ε, ποιότητα από τους γεωργούς, αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να τους κόβουμε και τα κονδύλια. Κάτι ακόμα που έλεγε η συγχύτρια ήταν να δώσουμε ένα, μια παραπάνω αξία και αυτό το είπε και προηγουμένω ο συνάδελφο στους επαγγελματίε γεωργού. γιατί δυστυχώς σήμερα με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν αποδίδουν πολύ. Πολλοί επενδυτές αγοράζουν τεράστιες εκτάσεις ε, το ανέφερε πριν ε, ο συνάδελφος για τη Γαλλία, αλλά και στην Ιταλία γίνεται το ίδιο. Και μετά αυτά, τα, αυτές τις εκτάσεις είτε τις καλλιεργούν ή τις υποκαλλιεργούν. Ακριβώς γιατί αυτός, οι μεγάλοι επενδυτές δεν θέλουν να φτιάξουν καλλιεργικά προϊόντα και να τα πουλήσουν, απλά θέλουν να έχουν γη που τους δίνει την συμβολή της ΚΑΠ εκτάριο. Αυτά, αυτή δεν είναι γεωργία, είναι επιχειρήσεις, είναι όμιλοι που στην ουσία διαχειρίζονται αυτά τα τεράστιες, τις τεράστιες εκτάσεις. Και εδώ λοιπόν πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τους επαγγελματίες γεωργούς και φυσικά την ποιότητα του προϊόντος. Και εδώ θεωρώ, γιατί εγώ παρακολούθησα λίγο το θέμα και στη Γεωργία και ο Τσιόλος συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό, ότι θα πρέπει να δούμε και την ανακατανομή των ταμείων, όχι μόνο ανά εκτάριο, ακριβώς για να αποφύγουμε την κερδοσκοπία, αλλά ανά εκτάριο, αλλά λαμβάνοντα υπόψη και άλλου δείκτε, όπω π.χ. την ποιότητα του γεωργικού προϊόντο, την εγκατάσταση τη ε, γεωργική εκμετάλλευση, αν είναι σε μια ορεινή περιοχή ο γεωργό ε, ε, καθαρίζει το νερό που χρησιμοποιεί ή καθαρίζει το, τις εκτάσεις του, τι χρησιμοποιεί ζυζανιοκτώνα ή όχι και τι ζυζανιοκτώνα. Α, λοιπόν, μια συμβολή, όχι μόνο ανά εκτάριο, γιατί αυτό οδηγεί στην κερδοσκοπή και το γνωρίζουμε όλοι, αλλά με βάση αυτό που παράγεται στο κάθε, στην κάθε έκταση, σε κάθε αγρόκτημα και πώς. Δηλαδή, να δίνουμε μια συμβολή αντίστοιχη με την ποιότητα. Και αυτό συμφωνεί και με τα όσα έλεγε η συγγέντρια. Δηλαδή, να ευνοήσουμε όσο γίνεται περισσότερο ένα ποιοτικό γεωργικό προϊόν, το οποίο θα ωφελεί και τον τελικό μας καταναλωτή, που είναι ο κεντρικός μας στόχος. Και εδώ συνδεόμενο Συνδεόμενη είναι η δυνατότητα να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τους γεωργούς στις δύσκολες περιοχές, στους λόφους και στα βουνά, όπου συχνά από τη στιγμή που εγκαταληφθούν, μένουν να καλλιέργεται, τα δάση καίγονται, γιατί από κάτω μένουν ένα-δυο μέτρα ε, υπόλοιπα η ξερά ε, ξερά στάχια ή έφλεκτα, εν πάση περιπτώσει, ξύλια, τελείως όμως απρόσεκτη με κίνδυνο μεγάλο πυρκαγιάς. Αν ήταν όμως πιο προσεγμένα τα εδάφια αυτά, δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και αυτό θα πρέπει να είναι λοιπόν μέσα στου στόχους μας. Το περιβάλλον, προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και υγεία, υγεία του τελικού καταναλωτή, αλλά και του γεωργού. Για να μην ξεχνάμε ότι όταν ο γεωργός ψεκάζει τα ζανιοκτώνα, τα αναπνέει κιόλα. Αν καταφέρουμε λοιπόν να πάμε σε έναν κόσμο πιο καθαρό και ταυτόχρονα βοηθήσουμε τον Γεωργό να χρησιμοποιήσει εναλλακτικέ μεθόδους, είναι καλό για τον καταναλωτή αλλά και για τον ίδιο τον Γεωργό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρώση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά μπορεί να πει κάποιος ε, για την κοινή πολιτική. Κάτι που μας εκπλήσει είναι ότι προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τη στρατηγική 2020 αλλά δεν ε, χρησιμοποιούμε τα πετούμενα μέσα από τον προϋπολογισμό για την κοινή γεωρική πολιτική. Αν θέλουμε να τονώσουμε την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, δεν μπορεί να τεράστιο κομμάτι του προϋπολογισμού να διατίθεται ε, στη Γεωργία όπως σήμερα. Θα ήθελα να, πάντως να κάνω πια κάποια ειδικότερα σχόλια για το περιβάλλον και πώς επηρεάζεται από τη γεωργία. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο αλλαγών, δηλαδή στον τομέα της γεωργίας. Μπορούμε ήδη να κάνουμε πολλά πράγματα και ήδη γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή κατευθύνουμε τις επιδότησεις προς τις καλλιεργητικές πρακτικές που ευνοούν το περιβάλλον. Επίσης διαλέγουμε τις ποικιλίε που καλλιεργούμε και κυκλοφορούν στην αγορά. Συζητούμε τη χρήση των παρασιτοκτών. προσπαθούμε να μειώσουμε τις ε, εκπομπές ε, κτλ. Ένα σωρό δράσεις, αλλά εγώ προσωπικά δεν ε, καταλαβαίνω πώς μπορούμε να αιτιολογήσουμε αυτό το φοβερό πόσο που δαπανούμε στην κοινή γεωργική πολιτική χωρίς να έχουμε άμεσο θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον. Ε, ε, αντιλαμβάνομαι ότι όλοι σκέφτονται το στομάχι τους, ε, καταλαβαίνω για ποιους λόγους διαμορφώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η κοινή γεωργική πολιτική, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ο φορολογούμενος ε, θα πρέπει να ε, πληρώνει τόσα λεφτά προς τους γεωργούς, ε, ενώ και εκείνο έχει ίδια δικαιώματα. Δεν μπορεί να πληρώνει ο φορολογούμενος για δημόσια αγαθά, για το ότι ζει ας πούμε στο φυσικό περιβάλλον, θα ήθελα να τονιστεί αυτό μέσα στην έκθεση. Είναι καλό σημείο εκκίνησης. Ελπίζω όμως να επανεστιάσουμε την προσοχή μας στα, στα ζητήματα που προανέφερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Ούσκι ζήτησε να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στα τσεχικά συνεχίζει μετά την πολωνική προσφώνηση του Πρόεδρου. Πίστευω ότι είναι σαφές από τη συζήτηση που έχει λάβει η χώρα ότι η κοινή αγροτική πολιτική όσο έχει αυτή τη στιγμή δεν είναι βιώσιμη. Η ΚΑΠ θα πρέπει να τροποποιηθεί. Είναι δύο πράγματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το ένα είναι η ανισοκατανομή των επιδοτήσεων για τη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας Τσέχος γεωργός παίρνει κατά μέσον όρο το 50% των επιδοτήσεων που παίρνει ένας γεωργός στα παλιά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο θέμα είναι το συνολικό τμήμα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 40% το οποίο κατα... καταναλώνεται στη γεωργία. Αν η Ευρώπη θέλει να είναι σε παγκόσμιο επίπεδο ανταγωνιστική, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να διατηρηθεί στο διηναικές και δεν έχει καν ηθικό χαρακτήρα. Καλό είναι να μιλάμε για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά θα πρέπει να κατανοήσετε τι κάνει η πολιτική μας με τις επιδοτήσεις στη γεωργία. Ως αποτέλεσμα αυτών των επιδοτήσεων καταστρέφεται η Αφρικανική γεωργία. Αυτά τα οποία υποτίθεται ότι κάνει δίνοντας με το ένα χέρι βοήθεια, τα καταστρέφει με το άλλο χέρι που δίνονται οι επιδοτήσεις. Αυτά τα χρήματα εξάλλου που δίνονται σαν βοήθεια πολλές φορές καταλήγουν στις τσέπες των Αφρικανών δικτατόρων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα προτείνω να υπάρξει κάποια ριζική λύση η οποία θα είχε αρνητικό αποτέλεσμα για το περιβάλλον και θα άφηνε την αγορά να τα αποφασίζει όλα και αυτό όπως είδαμε λειτουργήσε τα τελευταία 50 χρόνια για να δημιουργήσει ένα πλαίσιο διαστρεβλωμένο. Η προστασία λοιπόν του περιβάλλοντος, η προστασία του τοπίου και η ασφάλεια της ε, δημόσιας διατροφής όπως ελέγχθη προηγουμένω, αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της συζήτησής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Θέλω να ζητήσω από την Κομισιόν ο κύριος Σαντιάγο από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή Περιβάλλοντος καθώς και την κυρία Κάδεμπαρς ε, την ε, εισηγήτρια Ε, για το μέλλον της ε, κοινή ε, γεωργικής πολιτικής. Έχει μεγάλη σημασία ο δημόσιος διάλογος γιατί υπάρχουν μεγάλες εδαφικές προκλήσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος το περιβάλλον πλέον και λαμβάνεται περισσότερο υπόψη. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε στο δημόσιο διάλογο με αυτήν την έκθεση. Ποιοι είναι οι στόχοι της μεταρρύθμισης να είναι βιώσιμη η παραγωγή τροφίμων ενώ ταυτόχρονα να, ε, θα είναι βιώσιμη και η διαχείριση του περιβάλλοντος και να αναλαμβάνονται δράσεις ευνοϊκές για το περιβάλλον. Αυτή είναι η ουσία της προτινόμενης μεταρρύθμισης για να ευθυγραμμιστεί η κοινή γεωργική πολιτική με τη στρατηγική 2020. Είναι σαφές για μας ε, ότι ε, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις κοινή γεωργικής πολιτικής θα έχουν ιδιαίτερη σημασία στο μέλλον και όπως ε, αναφέρουμε και στο σχέδιο έκθεσης υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το πετύχουμε αυτό. Πρασινοποίηση των αμέσων ενισχύσεων στον πρώτο πυλώνα και δεύτερον κατευθύνοντας την ανάπτυξη της υπαίθρου προς την καινοτομία, προς την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την προστασία της υπαίθρου μεγαλύτερη πρασινοποίηση θα έχουμε τόσο ή άλλως ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί οι δράσεις καλύπτουν όλη την επικράτεια. Θα πρασινοποιήσουμε τους δύο πυλώνες και θα έχουμε περιβαλλοντικές δράσεις και στους δύο πυλώνες και τέλος θα βοηθήσουμε τους γεωργούς για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές οικονομικές προκλήσεις ενώ ταυτόχρονα θα τους βοηθούμε να αντέξουν στις περιβαλλοντικές πιέσεις. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ε, μιλήσαμε και για την απλούστευση τα μέτρα πρασινοποίησης ε, που θα εφαρμοστούν ε, στις άμεσες ενισχύσεις και στην ανάπτυξη υπαίθρου θα αναλυθούν, θα κάνουμε αξιολόγηση κόστος όφελος και φυσικά δεν θέλουμε να περιπλέξουμε το σύστημα, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις περιβαλλοντικές προκλήσεις στο μέλλον και πιστεύουμε ότι η πρασινοποίηση και η αλλαγή κατεύθυνση στην ανάπτυξη της υπαίθρου είναι ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά για να πάρουμε τις αποφάσεις μας θα περάσουμε από την αξιολόγηση αντικτύπου. Για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς υπάρχει μια αναφορά στο σχέδιο έκθεσης και στο προηγούμενο σημείο συζητήσαμε για αυτό το θέμα, δεν χρειάζεται τώρα να μπω σε λεπτομέρειες, δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα μέσω της κοινή γεωργικής πολιτικής Προφανώ προφανώς οι γεωργοί θα πρέπει να ε, εφαρμόζουν συγκεκριμένες διαδικασίες ούτως ώστε να λαμβάνουν μελλοντικώς ε, τις ενισχύσεις τους, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλες συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω και πάλι το λόγο στην κυρία Κάλιμπαχ για να κλείσουμε τη συζήτηση θέλω να ευχαριστήσω όλους οι οποίοι έλαβαν, χώρα, έλαβαν μέρος σε αυτή την ευρεία συζήτηση. Κάποιοι από αυτούς βέβαια που έλαβαν το λόγο δεν είναι παρόντες, οπότε πρέπει εγώ να ε, εστιάσω μόνο στους συναδέλφους οι οποίοι παραμένουν ακόμα στην αίθουσα. Ο στόχος μας λοιπόν είναι φυσικά πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε τη διατροφή των Ευρωπαίων, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία. Θέλουμε τη βιώσιμη γεωργία, θέλουμε να διατηρήσουμε τη βιοπικιλότητα και όπως θα πρέπει να μην παραγνωρίσουμε την ανάγκη να υπάρξει και μία έμεση τροποποίηση της χρήσης της γης και φυσικά να καταλάβουμε και ποιες είναι και οι επιπτώσεις της πολιτικής μας σε τρίτες χώρες. Θέλουμε να έχουμε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της κουλτούρας, του πολιτιστικού πλαισίου και την ε, διατήρηση των θέσεων απασχόλησης και να εξασφαλίσουμε μια ισοδίκαια πολιτική επιδοτήσεων. Επομένως, μια τέτοια πολιτική δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν έχουμε και την καλύτερη κατεύθυνση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Τώρα θέλω να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Δυστυχώς υπάρχουν στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τη δική μας αρμοδιότητα, όπως είναι παραγωγικά τα θέματα απλοποίησης της γεωργικής πολιτικής. Αυτά δεν μπορούμε εμείς να τα αντιμετωπίσουμε φυσικά στη γνωμοδότησή μας ως Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος. Και φυσικά Είμαι έτοιμη να συζητήσω μαζί σας για να συμπεριλάβω τις προτάσεις σας στην κοινή μας γνωμοδότηση. Και νομίζω ότι για αυτούς οι οποίοι είναι ακόμα στην αίθουσα, ό,τι είπανε το έχω απαντήσει. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 21η Μαρτίου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 12 Απριλίου. Στην Ολομέλεια τον Ιούνιο 2011. Εξαντλήσαμε την ημερήσια μας διάταξη, την πρωινή. Αν είναι ήδη εδώ οι συντονιστές, μπορούμε να περάσουμε αμέσως στη συνεδρίαση των συντονιστών. Αλλά μόλις που μου είπαν ότι στις 11.30 ε, είπαμε να έρθουν, άρα λοιπόν θα τα ξανα...